Äh, Εκτάκτο, σήμερα το απόγευμα έχουμε μικρή ακρόαση για ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα που είναι το μέλλον ε, της ευρωπαϊκής πολιτιστικής πρωτεύουσας. Είναι λίγο πρόωρο, αλλά δεν πειράζει να αρχίσουμε εγκαίρως, διότι κάποια στιγμή την Άνοιξη θα φέρει πρώτα πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ενδεχομένως να μπορούσαμε ήδη να επηρεάσουμε με τις ιδέες μας. Έχουμε στην Κριτική Επιτροπή δικά μας μέλη, έχουμε στείλει εμείς, έχουμε διορίσει εκεί, είναι τριετής η θητεία τους και μετά αποχωρούν. Έχουμε δύο εμπειρογνώμονες τώρα που ε, αποχωρούν, η κυρία Δόκτωρ Πλόντης και ο κύριος Δόκτωρ Βίζαν και επίσης έχουμε καλέσει και ένα ακόμα μέλος που δεν το στείλαμε εμείς Κάποιο άλλο το διόρισε, το Συμβούλιο μάλλον, αλλά είναι η πρώην συνάδελφο, η κυρία Ένικο Σόπκε, που ήταν και μέλο ε, τη Επιτροπή Πολιτισμού και χαιρόμαστε πραγματικά που έχουμε ενώπιον μα τρει πραγματικού εμπειρογνώμονε για την Ευρωπαϊκή Προσ... Πρωτεύουσα. Γνωρίζουμε ότι το 2019 λίγη η σημερινή μορφή το σημερινό πρόγραμμα και θα πρέπει να ε, μας προβληματίσει το μέλλον. Τι θα κάνουμε, θα συνεχίσει όπως έχει, κάθε χρόνο θα ορίζεται μία πόλη ή δύο περιφέρειες, τι θα γίνει. Ό,τι και να γίνει πολλές δυνατότητες και χαίρομαι που σήμερα έχουμε επισκέπτες από το Βελιγράδι, το οποίο Βελιγράδι καταβάλει προσπάθειες το 2020 να γίνει πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης. Όταν έχεις τέτοιους στόχους γνωρίζεις και γιατί εργάζεσαι. Το πρόβλημα είναι ότι δεν μπορούμε εμείς να το εγκρίνουμε έτσι. Ε, να ακούσετε, ε, ίσως να μάθετε και να κάνετε και την καλύτερη πρόταση. Λοιπόν, καλωσορίσατε όλοι και πάλι όσοι ενδιαφέρεστε. Δυστυχώς είναι πέμπτη απόγευμα, αλλά δεν είχαμε βρει άλλη ημερομηνία. Εμείς το θελήσαμε και εμείς θελήσαμε να μάθουμε από σας. Έχουμε τους τρεις εμπειρογνώμονες. Δέκα λεπτά έκαστος και λιγότερο, δεν χρειάζεται να τα εξαντλήσετε και μετά θα έχουμε και χρόνο να συζητήσουμε. Βεβαίω παρευρίσκεται εκτός αυτών και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο Γενικός Διευθυντής Σούχαν. που εργάζεται εδώ και πολύ καιρό σε αυτό το πρόγραμμα και παρευρίσκεται και ο κ. Κάμελ που γνωρίζουμε εδώ και καιρό επίσης για τα πολιτιστικά. Θα δώσω τώρα το λόγο στην κυρία Αγκλόντης. Παρακαλώ. Μπορείτε να μιλήσετε αγγλικά, γερμανικά, γαλλικά, ό,τι προερίστε. Αγγλικά. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που με διορίσατε ε, Ευρωπαία εμπειρογνώμονα. Τρεις φορές έχω διοριστεί με διαφορετική ιδιότητα κάθε φορά αλλά έτσι έγραψα και το διδακτορικό μου. Έκανα διδακτορική διατριβή για τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσε. Είναι ε, το πρώτο τέτοιο βιβλίο που γράφεται για αυτό το θέμα στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Συνεισφέρατε τα μάλα σε αυτή την προσπάθεια. Ε, γράφοντας λοιπόν αυτή τη διατριβή έκανα κάποια έρευνα και είχα αρκετό υλικό να εξετάσω 63 αιτήσει πόλεων έπρεπε να διαβάσω τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς και συνεντεύξεις. Um, και συμμετείχα βεβαίως και στην επιλογή και στην παρακολούθηση όλων των πρωτεύουσών το 2009 στο το 2013, που, 16 συγγνώμη, καταλαβαίνετε ότι είναι μεγάλη χρονική περίοδος. Και μετά από αυτή την έρευνα ε, και τις μελέτες μπορώ να θεωρήσω, μου επιτρέπετε ότι είμαι σε θέση να κάνω ορισμένες συστάσεις και να βγάλω ορισμένα συμπεράσματα. Τα προγράμματα έχουν βελτιωθεί ως προς την ποιότητά τους, ενώ ότι υποβολή υποψηφιωτήτων γνωρίζουν πλέον τα κριτήρια η πόλη και τη διαδικασία επιλογής, η οποία έχει καταστεί πιο διαφανής και πιο ε, σαφής. Υπάρχει μια διεθνής κριτική επιτροπή που μπορεί να εγγυηθεί και να διασφαλίσει ότι η ευρωπαϊκή διάσταση του προγράμματος προστατεύεται. Άλλος, υπάρχει ε, ένας πειρασμός, μια παγίδα να ε, θέλουν οι πόλεις να προχωρήσουν προς την οικονομική τους ανάπτυξη, όχι την πολιτιστική. Δηλαδή, αυτό που θα χρειαζόταν ίσως περισσότερη προσοχή είναι να γίνεται κατανοητή η ευρωπαϊκή διάσταση. Τι είναι αυτό το κριτήριο, τι είναι αυτή η έννοια. Χρειάζεται μεγαλύτερη διευκρίνηση. Αλλιώς, εκείνοι που προετοιμάζουν τις υποψηφιότητες θεωρούν ότι η ευρωπαϊκή διάσταση είναι να καλέσεις ξένους καλλιτέχνες στο φεστιβάλ σου ή στις συναυλίες. Όχι, δεν είναι αυτό η ευρωπαϊκή διάσταση. Είναι πολύ λίγος ο χώρος για την ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά και για τις ευρωπαϊκές προκλήσεις που έχουν να αντιμετωπίσουν. Και η Ευρώπη καθημερινά αντιμετωπίζει. Κάτι άλλο που κατέστη σαφέστατο μετά από όλα αυτά τα χρόνια είναι ότι η δράση της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Πρωτεύουσας είναι ο πιο μεγάλος τίτλος, ε, η μεγαλύτερη τιμή και το μεγαλύτερο κύρος που μπορεί να έχει μια πόλη. Και με όλη αυτή την κληρονομιά, με ό,τι σημαίνει αυτή η πολιτιστική πρωτεύουσα, αυτός ο τίτλος και η διάκριση θα πρέπει να συνεχιστεί. Θα πρέπει να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες για να διατηρηθεί η ευρωπαϊκή ανάπτυξη και η πολιτιστική ανάπτυξη αλλά το ανέφερα προηγουμένως αυτό. Τα προγράμματα και οι υποψηφιότητες θα πρέπει να έχουν μέσα τους ζωή, γιατί πολύ συχνά οι ντόπιοι πολιτικοί θέλουν να τα ρυθμίσουν όλα μόνοι τους, να τα αποφασίσουν όλα μόνοι τους και να τα επιβάλλουν στον κόσμο. Αυτού του είδους η διαδικασία είναι κατά της συμμετοχικής δημοκρατίας που εμείς αυτό θέλουμε να επικαλούμαστε και να προωθούμε όταν συνεργαζόμαστε και στην ε, Κριτική Επιτροπή. Η πόροι τώρα για την Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Πρωτεύουσα. Όποιο ασχολείται με αυτά τα θέματα και σε όποιον απευθύνθηκα εγώ, είχε εντονότατε επικρίσει. Και θα ήθελα να απευθύνω μια έκκληση προ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αυξηθεί η πρικοδότηση που αναφέρεται και δίνεται στο βραβείο Μελίνα Μερκούρη. Οι πόλεις επενδύουν πάρα πολύ για την ανάπτυξή τους στην κοινωνική συμπεριλήψη, βελτίωση της κατάστασης. Καλό θα ήταν να κάνει μια χειρονομία και η Ευρωπαϊκή Ένωση αυξάνοντας τα κονδύλια. Αν με ρωτήσετε αν θα πρέπει να συνεχιστεί η πολιτιστική πρωτεύουσα, βεβαίω και θα πρέπει. Δεν επιτρέπεται να τη σταματήσετε και να συνεχιστεί και να αναπτυχθεί έτσι περαιτέρω. Δεν υπάρχει καμιά άλλη πολιτιστική δράση στην Ευρώπη, έτσι με την ευρωπαϊκή σημαία, που να έχει τόση μεγάλη δυνατότητα να δημιουργεί τόσο ευρύ πεδίο και δίκτυο συνεργασία με τόσους πολλούς φορείς, από πολιτικούς φορείς, τοπικούς, περιφερειακούς, εθνικούς, διεθνείς, μέχρι και τον πολίτη της ίδιας της πόλης. Αυτό είναι πραγματικά κάτι το απίστευτο. Είναι ο μόνος διαγωνισμός όπου μπορούν να συμμετέχουν και πολιτικοί και κυβερνήσεις. Ακούστηκαν και κάποιες φωνές όταν προετοιμάζαμε τον νέο κανονισμό ότι ενδεχομένω καλό θα ήταν να περιορίσουμε τη δράση αυτή σε ορισμένε χώρε, μόνο στι μεγάλε χώρε, ίσω ξέρω εγώ. Και με ποια κριτήρια θα περιορίσει, θα αποκλείσει χώρε. Νομίζω ότι η διαδικασία θα πρέπει να παραμείνει όσο έχει σήμερα τόσο ανοιχτή, τόσο ευρεία. Όλες οι χώρες να έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν στο διαγωνισμό αυτό, ανεξαρτήτως μεγέθους ή της πολιτιστικής κληρονομιάς, της καλλιτεχνικής δυνατότητας, του δυναμικού, τη δημιουργικότητα. Κάθε χώρα έχει το δικαίωμα να κάνει μια τέτοια πρόταση. Εγώ δεν θα έκανα διάκριση με βάση το μέγεθος ή τη δυνατότητα μιας χώρας. Η διαδικασία τώρα της επιλογής. Υπάρχει μια επιτροπή που απαρτίζεται από διεθνεί εμπειρογνώμονε και θα πρέπει να συνεχίσει τι δραστηριότητέ τη, αλλά θα πρέπει να μα απασχολήσει και πάλι η δομή τη και η σύνθεση. Δηλαδή, η βέλτιστη λύση είναι να συνδυάζονται οι διεθνεί εμπειρογνώμονε με εθνικού, γιατί πολύ συχνά είχαμε την αίσθηση και πολλέ φορέ μα το έλεγαν και οι κυβερνήσει ότι στις χώρες τι ίδιε δεν υπάρχουν ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονε. άρα θα πρέπει να διορίσουν οι υπαλλήλου του Υπουργείου. Αν συμβαίνει κάτι τέτοιο, ειλικρινά εγώ προτείνω και προτιμώ να είναι διεθνής η Κριτική Επιτροπή, τελείω να αποφασίζει. Αλλά αυτό είναι για την επόμενη περίοδο. Μία πρόταση είναι αυτή. Πρόταση δεύτερη. Παρακαλώ, φροντίστε να υπάρχει ισορροπία στο φύλλο στην κριτική Επιτροπή. Οι γυναίκες είναι πολλές φορές μειονότητα και είναι δύσκολο να κάνουμε τη φωνή μας να ακουστεί. Και επίσης παρακαλώ να διατηρήσετε την ισορροπία της ηλικία. Είναι πολύ λίγοι νέοι στο πάνελ. Οι νέοι έχουν και αυτή πείρα. Και ένα τελευταίο, χωρί να είναι το λιγότερο σημαντικό, βεβαιωθείτε ότι τα νέα κράτη-μέλη εκπροσωπούνται στον ίδιο βαθμό με τα παλιά. Εγώ ήμουν η πρώτη που διορίστηκα από την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη και η μοναδική για πάρα πολλά χρόνια. Μπορείτε να το φανταστείτε. Εγώ τι ευθύνη φέρω στους ώμους μου. Was ε, very, very high. Ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Για δέκα χώρες εγώ αγωνιζόμουν και πάλευα. Λοιπόν, σας παρακαλώ, ε, ε, βεβαιωθείτε ότι θα είναι δεδομένη και ισορροπία μεταξύ παλιών και νέων κρατών μελών. Και μία τελευταία πρόταση και σχόλιο. Όταν λοιπόν συζητούμε για τα κριτήρια επιλογής ε, της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Πρωτεύουσα, μιλούμε και για την ευρωπαϊκή διάσταση που δεν ξέρουμε τι ακριβώς είναι, αλλά μπορούμε να το διευκρινίσουμε με τρόπο ώστε να αφορά σύγχρονες μορφές ανταλλαγής καλλιτεχνών Έχουμε τις πόλεις και τις πολίτες που αντανακλούν θαυμάσια τις φιλοδοξίες και των πολιτών και των πόλεων. Αλλά εγώ θα πρότεινα ένα ακόμα κριτήριο που θα αφορά τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στην πολιτική γειτονία και την εξωτερική πολιτική. Και αυτό είναι το κριτήριο της αλληλεγγύης. Η αλληλεγγύη είναι αξία. Δεν πρόκειται μόνο για την ένταξη και για την οικονομική ανάπτυξη. Η αλληλεγγύη είναι παγκόσμιο ιδανικό και την καταλαβαίνουν και οι πολίτες και στις πόλεις τις ίδιες, αλλά και είναι ένα ιδανικό και ιδεώδες που συμμερίζονται και η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Ηνωμένα Έθνη. Ακόμα και στους στόχους της χιλιετίας περί αλληλεγγύης πρόκειται ή στην πολιτική γειτονίας για ποιο λόγο δεν ζητούμε από τους πολίτες της Ευρώπης να συνεργαστούν μαζί μας, με τη στάση μας, τη δική σας, τη δική μας, του Κοινοβουλίου, για να προωθήσουν την ιδέα της αλληλεγγύης και να την γνωρίσουν μέσω της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Πρωτεύουσας. Ελπίζω να το συζητήσουν τα μέλη του Κοινοβουλίου και να το υιοθετήσουν αργότερα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για όλες τις προσπάθειες και την υποστήριξη που μας παρήχαν και σε μένα προσωπικά και στον Ανδρέα Βίσεντ. Κάποια στιγμή ξεπλάγει όλοι από την απήχηση που είχε αυτή η προσπάθεια. 16 υποψηφιότητε από την Ισπανία ήρθαν, 11 από την Πολωνία. Καταλαβαίνετε πόση δουλειά είχαν όλοι αυτοί για να προετοιμάσουν τις προτάσεις και τι υποψηφιότητες. Πρωτοφανής ήταν και... Θα ήθελα περισσότερη υποστήριξη και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο ανθρώπινο δυναμικό και στους οικονομικούς πόρους. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και για την ευκαιρία που μου δώσατε να είμαι Ευρωπαίοι εμπειρογνώμων και σας εύχομαι ότι καλύτερα. Σας ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος, και για το έργο σας. Το κάνατε γιατί εμείς σας το ζητήσαμε και για την ίδια σας τη σταδιοδρομία σας βοήθησε αυτό ακόμα καλύτερα. Θαυμάσια που βοηθούμε τον κόσμο να έχει καλύτερη σταδιοδρομία. Εργαζόμενοι για μας ταυτόχρονα. Ευχαριστώ. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Βίσεν. Παρακαλώ. Uh, Σα ευχαριστώ πολύ και καλησπέρα σε όλου. Ε, θα μιλήσω στα αγγλικά, οπότε μπορείτε ίσω άμεσα να με καταλάβετε όλοι. Proves Την πρώτη φορά που ήρθα εδώ στην Επιτροπή Πολιτισμού ήταν πριν από 20 χρόνια. μέσα στα πλαίσια του Ινστιτούτου ΕΡΙΚΑΤ. Τότε η συνεδρίαση και όλα τα σχετικά ήταν κάπως προσωρινά. Η θέση του πολιτισμού στα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν πολύ ευάλωτη Από τότε πολύ προχωρήσαμε και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Ινστιτούτο μας. Ο ε, ρόλος της Επιτροπής ήταν πάρα πολύ σημαντικό για να δοθεί ε, ο πολιτισμός ε, στην... να βρεθεί ο πολιτισμός στο σωστό του ρόλο και η ΕΚΟΚ βέβαια ήταν πάρα πάρα πολύ σημαντική εδώ. Και εμείς όμως προχωρήσαμε στο Ινστιτούτο μας. Πριν από 8 χρόνια δημοσίευσαμε τη μελέτη Δημιουργική Ευρώπη με την βοήθεια κάποιων ιδρυμάτων ευρωπαϊκών και χαίρομαι που τώρα επέλεξε η Κομισιόν τον ίδιο τίτλο για το δικό της πρόγραμμα. Επίσης είχαμε μία μελέτη για τους ε, καλλιτέχνες στην Ευρώπη. Μετά προετοιμάσαμε μία μελέτη για το Ευρωπαϊκό Έτος ε, Διαπολιτιστικού Διαλόγου του 2008. Είμαι σίγουρος ότι πολλά θα μπορούσαν ε, να ακολουθήσουν και θα ακολουθήσουν. Τώρα θα αναφερθώ στην εμπειρία μου. Έχετε ένα φυλάδιο στα χέρια σας. Από όσοι κατάλαβα, έχει μοιραστεί σε όλους, δεν χρειάζεται να σας τα διαβάσω όλα αυτά. Μπορείτε να διαβάσετε μόνοι σας τις λεπτομέρειες. Πρέπει να τονίσω ότι αυτό δεν είναι μια γενική ε, εικόνα, όπως είπε η Δανούτα, για όλα τα θέματα, αλλά αναφέρονται ορισμένα τα προβλήματα που αντιμετώπισα εγώ ως μέλος αυτής της Κριτικής Επιτροπής. που ήμουνα κάπως ε, εκείνος που έβλεπε τα πράγματα απ' έξω, γιατί δεν ήμουν ποτέ υπεύθυνο για κάποια πολιτιστική πρωτεύουσα ή οτιδήποτε άλλο. Η εμπειρία μου είναι μια εμπειρική αξιολόγηση και όπως είπε και η Τανούτα έχω και εγώ να πω ότι πολλά μπόρεσα να μάθω σχετικά με το συγκεκριμένο αυτό πρόβλημα. Ορισμένα από αυτά που θέλω να τονίσω απορρέουν από αυτή την εμπειρία. Ορισμένα τα ανέφερε η Δανούτα. Είναι περίεργο να βλέπει κανένα πώ ερμηνεύονται τα προγράμματα διαφορετικά από κάθε χώρα. Ορισμένες υποψήφιες θεωρούν ότι αν είναι τμήμα ενός ευρωπαϊκού δικτύου, φτάνει. Αυτό βέβαια δεν είναι πολύ ικανοποιητικό και θα ήταν καλό να έχουμε περισσότερες διευκρινήσεις. Έχω όμως μια συγκεκριμένη εικόνα και δεν ε, διστάζουμε να ανταλλάσσουμε τις διαφορετικές μας απόψεις. Η θέση μου λοιπόν είναι ότι πιστεύω ότι εκτό από συγκεκριμένα κριτήρια που πρέπει να πληρούν όλοι οι υποψήφοι, θα πρέπει να έχουμε κατά νου όλη τη διαδικασία ΕΚΟΚ. Και από τη διαδικασία αυτή θα πρέπει να απορρέει η ποικιλομορφία. Δηλαδή, κατά τη γνώμη μου, οι διάφορες ε, πόλεις θα πρέπει να έχουν και κάποια διακριτικά στοιχεία δεν είναι χρήσιμο όλες να κινούνται πάνω στο ίδιο ευρωπαϊκό πρόγραμμα που να είναι το ίδιο παντού. Θα πρέπει να έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της ε, περιφέρειας, της ε, πόλης που είναι υποψήφια. Ορισμένες φορές αυτό δεν ήταν πολύ ξεκάθαρο. Επίσης, Μάθαμε διάφορα από τα αποτελέσματα της πρόσφατης μεταρρύθμισης. Και όπως είπαμε είναι δύσκολο να αξιολογηθούν 16, 16 υποψηφιότητες αν έχει κανένα μονάχα μισή ώρα παρουσίαση στον πρώτο γύρο και άλλη μισή ώρα αργότερα. Αυτό δεν αρκεί για να αξιολογηθούν το έργο αυτών των υποψηφίων για να δουν κανένα αν έχουν πραγματικές ευκαιρίες, εάν πραγματικά πληρούν τους στόχους του προγράμματος. Ανησυχώ, γιατί σε κάποιες από αυτές τις προσφορές παίζουν ένα ρόλο και άλλα θέματα, παραδείγματος χάρη η οικοδόμηση μεγάλων υποδομών, αεροδρόμια, δρόμοι κλπ. που αποκτούν όσο πάει και μεγαλύτερη σημασία. Γιατί είπαν εντάξει, αν τελικά κερδίσει κανένα, θα είναι πιο εύκολο να πραγματοποιήσουμε τα έργα αυτά. Είναι φυσικό να σκέφτεται κανένα έτσι, αλλά το πρόγραμμα δεν είχε αυτό το στόχο ποτέ για την ε, ανάπτυξη αυτής της υποδομής. Ίσως αυτό να μπορέσει να είναι ο καρπός μιας επιτυχούς υποψηφιότητας, αλλά δεν θα πρέπει να είναι ο κύριος στόχος της υποψηφιότητας. Η διαφορά που υπάρχει μεταξύ των φτωχών και των πλουσίων χωρών ή πόλεων αναφέρθηκε ήδη. Και νομίζω ότι θα μπορούσε κανένας να προσπαθήσει να βρει έναν ευφυή μηχανισμό διάκρισης για αυτές τις διαφορές. το ίσως το οικονομικό υπόβαθρο που είναι πάρα πολύ διαφοροποιημένα μεταξύ των διαφόρων υποψηφίων και να υπάρχει ένας τρόπος ενίσχυσης εκείνων που έχουν λιγότερους πόρους. Ήδη ίσως στη φάση της υποψηφιότητας. Γιατί ας είμαστε ειλικρινείς, ορισμένες από τις πόλεις αυτές πανούν ήδη πολλά στην προετοιμασία της υποψηφιότητάς τους. Και αυτό κατά κάποιον τρόπο εξαφανίζεται το χρήμα, κερδίσουν και ίσως μάλιστα θα δαπανηθούν τα χρήματα αυτά και δεν μπορούν να αναπτυχθούν άλλες σημαντικές πολιτιστικές επενδύσεις σε τοπικό επίπεδο. Όσον αφορά τώρα την ε, διαδικασία και τη σύνθεση των πάνελ, αναφέρα στο έγγραφό μου πόσο σημαντική είναι η ανεξαρτησία του πάνελ αυτού. Ίσως θα υπάρχουν πιο έντονες δεσμεύσεις στο μέλλον ή θεωρήσουμε ότι η ανεξαρτησία δεν μπορεί να επιτευχθεί πλήρως. Εγώ θα προτιμούσα όμως η σύνθεση να μην προσανατολίζεται τόσο προς τα κράτη όπως το είδαμε σε ορισμένε φορές. Και εδώ συμφωνώ με την Τανούτα. Και όταν είχαμε τόσους πολλούς υποψήφιους ήταν δύσκολο να βρούμε τις σωστές διαδικασίες ψηφοφορία. Στα τελευταία χρόνια αλλάξαμε πολλές φορές την μέθοδο ψηφοφορίας. Συλλέξαμε βέβαια εμπειρίες, πάντα καταφέραμε τελικά να συμφωνήσουμε, αλλά θα ήταν ίσως καλύτερο να υπάρχουν διαδικασίες ψηφοφορίας που να λαμβάνουν υπόψη αυτές τις διαφορετικές ε, προϋποθέσεις. Πιο εύκολο να διαλέξει κανένα μεταξύ 2 ή μεταξύ 15. 15 είναι πολύ δύσκολο, 2 είναι εύκολο. Το τελευταίο σημείο, και αυτό είναι το σημαντικότερο για μένα, γι' αυτό κάνω εγώ. Η έρευνα και ανάπτυξη κριτηρίων αξιολόγησης, εδώ και 30 χρόνια κάνω αυτή τη δουλειά. Και έχω την εντύπωση ότι η μία αξιολόγηση εξ των πρωτοβουσών Δηλαδή αξιολόγηση το τι έκαναν οι πόλεις αυτές και ποιο ήταν το αποτέλεσμα των προσπαθειών τους, αυτή η αξιολόγηση έχει προχωρήσει πολύ και ακολουθεί στάνταρ διαδικασίες παντού. Αλλά δεν ισχύει το ίδιο όσον αφορά την εξάντε ε, αξιολόγηση, όσον αφορά τις υποψηφίες δηλαδή οι πόλεις. Είναι πολύ δύσκολο να αξιολογήσει ένα τόσο μικρό πάνελ αυτές τις υποψηφιότητες και να δει κατά πόσον παραβλέπετε κάτι ή αν πραγματικά είναι σύμφωνα με τους δύο κύριους όρους για την υποψηφιότητα, θα ήταν καλό τα κριτήρια αυτά να μπορούν να εξολογηθούν εκ των προτέρων για να μπορέσει το πάνελ να βασιστεί σε αντικειμενικά στοιχεία. Όχι μόνο δηλαδή στην ίδια την ε, πρόταση της ε, Νογοπόλης αυτά θα πρέπει να εξαρτηθούν, θα πρέπει να εξαρθεί το δυναμικό της πολιτιστικά της πόλης αυτής, το προφίλ και τη δυνατότητα από οικονομική πλευρά να πραγματοποιηθεί η πρόταση αυτή. Εγώ μόλι ήρθα από μια συνεδρίαση που είχαμε χτες που ελέγξαμε κάποιε πρωτεύουσε και πάλι είχαμε αυτή την κατάσταση που είχαμε ξαναδεί στο παρελθόν. Ότι κονδύλια που τους είχαν υποσχεθεί εξαφανίστηκαν ξαφνικά. Όλο το θέμα λοιπόν που ήταν πάρα πολύ σημαντικό για μας και για το οποίο εμείς δώσαμε τον τίτλο σε αυτή την πόλη χάθηκε ξαφνικά γιατί δεν υπήρχαν τα χρήματα να χρηματοδοτηθεί αυτή η δράση και θα πρέπει να δούμε ποιος είναι τελικά υπεύθυνο για την διαχείριση της διαδικασίας και να εξετάσουμε κατά πόσο εκτός από τις υποσχέσεις που υπάρχουν ε, οι χώρες παίζουν το σωστό ρόλο ή τι πρέπει να γίνει για να εξασφαλιστεί καλύτερα ότι αυτά που έχουν εγγραφεί στην υποψηφιότητα, στο έγγραφο της υποψηφιότητας, μπορούν να τηρηθούν και δεν εξαφανίζονται μετά από μερικούς μήνες. Αυτέ είναι ορισμένε από τι εμπειρίε που δεν θέλω να σα παρουσιάσω και ευχαριστώ να συζητήσω μαζί σα. Ευχαριστώ πολύ. Πρώτα εγώ σα ευχαριστώ κύριε Βίζαντ. Θα δώσω το λόγο στη φίλη Ενίκο Σίπσκε που ήταν υπουργό ε, πολιτισμού στο Λουξεμβούργο και είχε την υποψιότητα δύο φορέ. Δύο φορέ δεν ήτανε? Ναι, δύο. Θα μιλήσω γαλλικά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ο θεσμός των πολιτικών πρωτευουσών είναι ένα από τα πιο πετυχημένα προγράμματα και πρόκειται για ένα από τα προγράμματα τα οποία έδωσαν μεγαλύτερη ορατότητα στις πολιτιστικές μας πολιτικές. Τώρα ήρθε η ώρα να προβληματιστούμε για το μέλλον αυτού του προγράμματος, διότι πρέπει να ξαναδούμε τον τρόπο επιλογής ε, δεδομένης της κεκτημένης εμπειρία. Και εγώ, κυρία Πρόεδρε, θα κάνω μία αναδρομή της ε, εμπειρίας μου, της επαγγελματικής μου εμπειρίας. Εγώ πρώτα συμμετείχα στο Συμβούλιο, για μερικά χρόνια, μετά ήμουν ευρωβουλευτής για μία θητεία και σήμερα από το, και από το 2006 ασχολούμαι με αυτό το θέμα και μπόρεσα να παρακολουθήσω όλη τη διαδρομή μέσα από τους διοικητικούς με άνδρους όλης αυτής της ιστορίας. Το 2002 ήμουνα ακόμα υπουργό όταν χρειάστηκε να αποφασίσουμε για την πρωτεύουσα του 2009 στο Λουξεμβούργο. Στο Συμβούλιο Υπουργών είχαμε καταρχήν την απόφαση με ομοφωνία που δημιούργησε πρόβλημα. Όπως επίσης και για το 2000 είχαμε 9 προτάσεις και ο μόνος τρόπος για να λύσουμε το πρόβλημα ήταν να ορίσουμε όλες τις πρωτεύουσε και τις εννέα πόλεις δηλαδή και δεν είχαμε ορατότητα. Χρειάστηκε πολλή διπλωματία και πολλές διαπραγματεύσεις στο Συμβούλιο για να πείσουμε έναν Υπουργό να αποσύρει το όνομα το οποίο είχε προτείνει οι προσδοκίες και η πίεση σε εθνικό επίπεδο ήταν μια σημαντική πολιτική πρόκληση. Τώρα από το 2000 μέχρι για το 2019 είπαμε ότι κάθε χώρα θα πρέπει να ορίζει μία πόλη κατά προαίρεση και πρόκειται για μία απόφαση που είχε ληφθεί από 15 μέλη πριν από τη διεύρυνση. Το 85 όταν υποβλήθηκε η πρόταση συνοδευόταν και από πολύ σημαντικές προτάσεις τις οποίες δεν ασχολήθηκε ποτέ κανένας να τις εφαρμόσει. Έχουμε λοιπόν το πρώτο ψήφισμα του 85 το οποίο αναφέρει τη συνεισφορά των κρατών μελών στα, στα πλαίσια της επιλαγμένης πόλης. Αυτό θα είχε δώσει όμως μια ευρωπαϊκή διάσταση εξασφαλισμένη, δηλαδή μία πρωτεύουσα, πολιτιστική πρωτεύουσα σε κάθε κράτος μέλος και που θα ήταν χρηματοδημένη από το κράτος μέλος θα μπορούσαμε να προβάλλουμε την ευρωπαϊκή κουλτούρα της κάθε πόλης που θα ήταν πρωτεύουσα. Υπάρχουν όμως και διαρθωτικά διαρθρωτικά προβλήματα, γιατί υφίστανται σε όλες τις χώρες μας. Τις περισσότερες φορές είναι τα Υπουργεία Εξωτερικών που ασχολούνται με την πρόθεση της εθνικής, ε, του εθνικού πολιτισμού στο εξωτερικό. Υπάρχουν λοιπόν δικέφαλες ε, διαρθρώσεις καταμερισμένη σε πολλά υπουργεία, των οποίων η δράση εκεί αποτελεσματικότητα έχει να κάνει με επικάλυψη αρμοδιοτήτων, αλλά επίσης και με περιορισμένα μέσα στη διάθεσή τους για να προωθήσουν την εξαγωγή του πολιτισμού. Αυτό το ωραίο όραμα για την Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Πόλη, που μετά την ονομάσαμε πρωτεύουσα, δεν την εκμεταλλευτήκαμε σωστά θα χρειαζόταν κάτι τέτοιο, θα έπρεπε κάτι τέτοιο να γίνει ένα πραγματικά μοντέλο κινητικότητας, ε, συμμετοχής ε. και θα έπρεπε να συμβάλλει και στη σχέση μεταξύ των κρατών μελών. Οι αδυναμίες ε, σε εθνικό επίπεδο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα μπορούσαν να μας οδηγήσουν στο να δημιουργήσουμε ένα think tank για όλες τις πολιτικές με προβλήματα, όπως εκείνες της ολοκλήρωσης ή της πρόληψης των συγκρούσεων κλπ. Δεν θα έπρεπε λοιπόν εμείς να θεωρούμε τον πολιτισμό ως ένα άθροισμα όλων των φεστιβάλ, των παλέτων, των ορχιστρών ή των ε, οπερών θα έπρεπε να έχουμε ένα σχέδιο ηθικής ανοικοδόμησης σε μία περίοδο απελπισίας και παρακμής. Θα έπρεπε να <coughs> δημιουργήσουμε ένα νέο κίνητρο για την δημιουργικότητα. Υπό αυτή την πλευρά λοιπόν η πολιτιστική πρωτεύουσα θα έπρεπε να εκμεταλλευτεί αυτή τη δημοτικότητα και να βρει μια νέα πνοή μετά από το 2019. Λοιπόν, το 1995 το Λουξεμβούργο ήταν πρωτεύουσα όλων των πολιτισμών. Το πρόγραμμα είχε ετοιμαστεί από τον προκάτοχό μου, τον Ζακ Σαντέρ. Και η εμπειρία μου θα, αυτά που θα σας πω δηλαδή θα σας σοκάρουν ίσως αλλά θα έπρεπε να υπάρχει μία διάκριση μεταξύ των διαφόρων παραγόντων. Θα έπρεπε να εμπλακούν και οι πολιτικοί. Είχαμε μία διαχειριστική επιτροπή στο Λουξεμβούργο συμμετείχε ο, η Δήμαρχος, ο υπουργό, Υπουργός Πολιτισμού, οι υπάλληλοι του Δήμου, <coughs> οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι το Υπουργείο Οικονομικών και εγώ από αυτήν την ομάδα έμαθα να αντιμετωπίζω τα πρακτικά προβλήματα, αλλά μέσα από τη συλλογική συζήτηση το σχέδιο ευόδωσε. Εγώ δεν είμαι βέβαιη ότι αν βγάλουμε από τη μέση τους πολιτικούς θα, θα, θα μπορέσουν να συνειδητοποιήσουν ε, το τι παίζεται. Η ελευθερία έκφρασης είναι σίγουρα η βασική αρχή που πρέπει να σεβαστούμε. Εγώ θα ήμουν αντίθετη να, να δεχθώ οδηγίες ε, για τον διορισμό του προϊσταμένου της ομάδας. Εγώ έχω μόνο την Κομισιό να σεβαστώ. Όσον αφορά στον προϋπολογισμό, Πρέπει να σας πω το Λουξεμβούργο τον καιρό, τον καιρό εκείνο ήταν υπανάπτυκτο. Μετά από την κρίση του, του, στο Χάλιβα του 82 η κυβέρνηση ξανά φτιαχνε από την αρχή <coughs> τους, ε, τον εθνικό προϋπολογισμό. Αλλά για να μπορέσουμε να καλύψουμε το κενό στήσαμε μία μεγάλη ε, τέντα για όλη τη χρονιά όπου είχαμε εκδηλώσεις. Και ο κόσμος πίστηκε ότι οι πολιτιστικές υποδομές είναι χρήσιμες. Εγώ δεν θέλω να πιέσουμε ιδιαίτερα στο θέμα των υποδομών. Και η τάση αυτή επέτρεψε, το να, η τάση να επιβάλλουμε στις υποψήφιες χώρες να οι πόλεις να επενδύσουν στον τομέα αυτό είναι ένα δίκοπο μαχαίρι υπάρχει το καλό να πιστούν ότι ναι, χωρίς πολιτιστική υποδομή δεν υπάρχει δυνατότητα πολιτιστικής ανάπτυξης. Η επιβολή όμως των επενδύσεων θα πρέπει να συνδέεται με την εθνική κατάσταση. Και θα πρέπει κάθε φορά που, μια, που δημιουργείται μια υποδομή να βάζουμε και μια αναμνηστική πλάκα που να θυμίζει ότι φτιάχτηκε επ' ευκαιρία της πολιτιστικής πρωτεύουσας. Όλα αυτά λοιπόν ήταν επιτυχία για το Λουξεμβούργο και το 2007 χρειάστηκε να προβληματιστούμε γύρω από ένα άλλο πρόγραμμα όπου χρειάστηκε να έχουμε ένα διασυνοριακό πρόγραμμα. Έπρεπε να παρουσιάσουμε το πρόγραμμα αυτό το 2002. Είχαμε την επιλογή μιας εταιρικής πόλης για ένα μήνα και κράτησε μετά ένα χρόνο. Και επιλέξαμε το Σιμπίου στη Ρουμανία, όταν ακόμη αυτή η χώρα δεν ήταν μέλος. Αυτή η συνεργασία ήταν πάρα πολύ σημαντική και είχαμε αηφόρο συνεργασία μεταξύ των, των πόλεων. Και για το Σιμπίου <coughs> ήταν μια μεγάλη τύχη διότι με το, τωρινό σύστημα αυτή η πόλη δεν θα οριζόταν ποτέ ως πολιτιστική πρωτεύουσα. Το Λουξεμβούργο επίσης εκμεταλλεύθηκε αυτόν τον ορισμό ως πρωτεύουσα για να μπορέσει να προωθήσει αυτό το πολιτιστικό μοντέλο διασυνοριακής συνεργασίας. Η ευρύτερη περιοχή της ε, ΣΑΡ του ΛΟΡ και του Λουξεμβούργου δημιουργήθηκε μέσα από έναν στενό οικονομικό δεσμό που είχαμε στο παρελθόν. Και εμείς ανασύραμε ένα δίδαγμα από αυτό, συμπεριλαμβάνοντας ένα συνολικό πρόγραμμα. Τώρα, η, η κριτική επιτροπή που ασχολήθηκε με την επιλογή δεν γνώριζε την ευρύτερη, ε, την ευρύτερη περιοχή. Αλλά έτσι όπως υπάρχει εδώ και δεκαετίες, δηλαδή με τη διακοινοβουλευτική αντιπροσωπεία και με τις υπουργικές συνδετήσεις. <coughs> Εγώ θεώρησα τότε ότι θα έπρεπε να είχαμε ένα ευρωπαϊκό, ε, μια ευρωπαϊκή κριτική επιτροπή. διότι φοβόμουν ότι οι αποτυχίες θα ριχνόντουσαν στην πλάτη της Κομισιόν και της Ευρώπης. Θεώρησα λοιπόν ότι θα έπρεπε με τη σειρά να διαλέγει το Συμβούλιο. Με την εμπειρία που είχαμε όμως σήμερα με την Ισπανία και την Πολωνία όπου είχαμε πάρα πολλούς υποψήφιους και προγράμματα δύσκολο να επιλέξουμε δεν θα μπορούσαμε να φανταστούμε έναν διαγωνισμό σε εσωτερικό επίπεδο. Θα έπρεπε λοιπόν εμείς να εκμεταλλευτούμε όλες τις υποψήφιες πόλεις που θα πρέπει να επεξεργαστούν το πρόγραμμα για να παρουσιάσουν την υποψηφιότητά τους. Η απαγοήτευση βέβαια δεν είναι πάντοτε το καλύτερο, ο καλύτερος σύμβουλος. Τώρα όμως πρέπει να δούμε Πώς θα ορίζουμε τον καλύτερο, η Ευρωπαϊκή Κριτική Επιτροπή είναι η καλύτερη, δεν δέχεται πιέσεις. Και πρέπει εδώ να πω ότι η Κομισιόν κάνει ό,τι μπορεί για να προστατεύσει τα μέλη της, της Επιτροπής Επιλογής από οποιαδήποτε πίεση. Θα πρέπει να υπογράφουν ε, μία δήλωση για το ασυμβίβαστο, θα πρέπει να μην κάνουν δηλώσεις στον τύπο, και να μην κάνουν τίποτα δημοσίως χωρίς τη συμφωνία της Κομισιόν. Η μελέτη γίνεται με, σύμφωνα με τις... Ε, η επιλογή συγγνώμη, γίνεται σύμφωνα με τις μελέτες οι οποίες στέλνονται κατοίκων στους υποψήφιους <coughs> κατοίκων συγγνώμη στην <coughs> Επιτροπή που επιλέγει τα κράτη. Και όλα αυτά γίνονται ανεξάρτητα και μπορούμε να παρακολουθούμε από την αρχή ως το τέλος την επιλογή. Θα έπρεπε <coughs> να παρακολουθούμε ενιαία την κάθε προτινόμενη πόλη. Τα μέλη της Επιτροπής ε, θα πρέπει να επισκέπτονται και να ε, δημιουργούν και προσωπική εμπειρία για την κάθε πόλη. Να υπάρχει μία σχέση εμπιστοσύνης, πολλές φορές η επίσκεψη επιτόπου μας βοηθάει να ξεμπλοκάρουμε εγκλωβισμένες καταστάσεις και οι υποψήφοι ίδιοι λένε ότι η βοήθεια της Επιτροπής τους είναι πολύτιμη. Όμως, η έλλειψη επαφών με τις άλλες πολιτιστικές πρωτεύουσες δεν είναι καλό πράγμα. Χρειάζεται λοιπόν να έχουμε ένα δίκτυο των παλαιών πρωτεύουσών, πολιτιστικών πρωτεύουσών, <coughs> και να μπορούν δηλαδή να συνεχίζουν και μετά από τη χρονιά που είναι πολιτιστικές πρωτεύουσες στενή συνεργασία να βοηθούν κατά την προπαρασκευή των νέων, κατά την προετοιμασία των νέων υποψηφίων με συμβουλές. Στα πανεπιστήμια όμως υπάρχει ένα τέτοιο δίκτυο των πολιτιστικών πρωτεύουσών Δηλαδή οι πολιτιστικές πρωτεύουσες ε, έχουν ένα δίκτυο σε επίπεδο πανεπιστημίων. Το τοπικό στοιχείο επίσης θα πρέπει να τονιστεί. Είναι πολύ καλό το μιλάμε εμείς για ευρωπαϊκή διάσταση. Αλλά από την άλλη μεριά ο κόσμος δεν θα πρέπει να έχει την εντύπωση ότι τους επιβάλλεται ένα σχέδιο και ότι το πιλοτάρουν εξωτερικοί παράγοντες. Όλα αυτά δεν γίνονται από τη μία μέρα στην άλλη. Το να καλεί κανείς εμπειρογνώμονες είναι πολύ σημαντικό, αλλά θα έπρεπε όμως να δημιουργηθούν και περίοδοι άσκησης στάζ στις χώρες που είναι υποψήφιες για να μπορούν να καταρτίζονται οι ομάδες. Το σημερινό μοντέλο έτσι όπως λειτουργεί βρίσκεται υπό την επιρροή της Κομισιόν και ο προϋπολογισμός είναι αυτός που είναι και ο χρόνος εργασίας δεν επιτρέπει ιδιαίτερο προβληματισμό και συζήτηση. Η Επιτροπή Επιλογής θα πρέπει να αναλάβει <coughs> μόνο την ευθύνη της επιλογής, χωρίς παρέμβαση ή βοήθεια προς τους υποψήφιους. Κοιτάστε, πρόκειται για το πρόγραμμα φάρο όλων των πολιτιστικών προγραμμάτων. Θα έπρεπε αυτό το πρόγραμμα να έχει πιο αηφόρες επιπτώσεις και να λειτουργεί ως μοφλό. Συμπεράσματα. Θα πρέπει να έχουμε ένα αηφόρο σχέδιο πολιτιστικής ανάπτυξης που να επικρατεί επί των προγραμμάτων εκδήλωσης, να είναι κάτι πιο σταθερό, να γίνεται μία αξιολόγηση των επενδύσεων, να έχουμε τα να, να ενσωματώνουμε σχολικά προγράμματα, πολιτιστικές τεχνικές, να μπορούμε να ενσωματώνουμε ε, ιδιομορφίες τοπικές ε, και μειονότητες. Θα πρέπει να έχουμε ένα δίκτυο των παλαιών ε, πολιτιστικών πρωτεύουσών. Θα είχαμε 12 πρωτεύουσες έτσι με κυκλική προεδρία που θα μπορούσαν να είναι ένα φόρουμ. Επίσης θα έπρεπε επίσης να λύσουμε σε ένα γενικότερο πλαίσιο το θέμα της κινητικότητας των καλλιτεχνών και να ξεπεράσουμε όλα τα εμπόδια τα οποία υφίστανται στην κινητικότητα των καλλιτεχνών θέτοντας σε πράξη όσα υπαγορεύει η έκθεσή σας σχετικά και που εμποδίζονται όχι από τους ε, Υπουργούς Πολιτισμών αλλά από άλλους υπουργούς που ασχολούνται με τις ε, πολιτικές για τις θεωρήσεις ε, με τα οικονομικά. Θα ήθελα λοιπόν το Κοινοβούλιο να δώσει σαφείς κατευθύνσεις σε ορισμένους τομείς και να παλέψει ούτω ώστε ο πολιτισμός να λάβει τη θέση που, ε, που του αρμόζει. Κύριε Φίσας. Ευχαριστώ Πρόεδρε, νομίζω ότι είναι ένα θέμα πραγματικά σημαντικό. Αλλά εγώ έχω ορισμένε αμφιβολίες. Πρώτα απ' όλα για το σύστημα επιλογής Εάν κατάλαβα καλά, από το 2016 τα κράτη-μέλη θα προτείνουν την πόλη. Οπότε δεν ξέρω εγώ ποιος είναι αλήθεια ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή της Κομισιόν. Διότι δύσκολο είναι να πει κανείς όχι στην πρόταση που έχει υποβάλει ένα κράτος μέλος. Υπήρξαν διάφορα συστήματα εγώ θα ήθελα να ξέρω ποιο είναι το πιο ενδιαφέρον από όλα. Και επίσης θα ήθελα να ξέρω αν η επιλογή γίνεται πραγματικά για πολιτιστικούς λόγους ή αν επηρεάζεται από πολιτικούς λόγους. Επίσης υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο σχέδιο, ε, κάποιο συγκεκριμένος απολογισμός για το τι επιπτώσεις ε, ε, οικονομικά, στον οικονομικό και τουριστικό τομέα έχουν οι πολιτιστικές πρωτεύουσες. Κυρία Τρέπε. Ευχαριστώ τον εμπειρογνώμονα μας. Ε, πολύ ενδιαφέρουσες ε, οι συστάσεις και τα συμπεράσματα σας. Έχω κάποια ερωτήματα προς την Τανούτα Γλόντες, γιατί αυτό που είπατε εσείς είναι ότι ο βιομηχανικός τομέας που απασχολεί εκατομμύρια ε, Ευρωπαίων πολιτών θα πρέπει να έχει τις ίδιες δυνατότητες ανάπτυξης όπως και άλλοι τομείς. Τι εννοούσατε όσον αφορά μέσα προϋπολογισμό κλπ. Τι είχατε κατά νου. Μετά αναφέρεστε στην εισαγωγή ενό ευρωπαϊκού πολιτιστικού μήνα σε τρίτες χώρες. Τι έχετε κατά νου, πώς θα λειτουργούσε κάτι τέτοιο. Μ' άρεσε επίσης που είπατε ότι θα θέλατε παντού να υπάρχει ε, κάθε χρόνο συγγνώμη, δεν τα μπέρδεψα λιγάκι κάθε χρόνο να υπάρχει συνεργασία μεταξύ μιας ανατολικής και μιας δυτικής πολιτιστικής πρωτεύουσας. Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να συμμετάσχω στη συζήτηση. Κάτι που είπε ο κ. Βίλαν δεν θέλω να το δεχτώ έτσι. Δεν νομίζω ότι ο ανταγωνισμός μέσα σε μια χώρα είναι παράλογος γιατί στο τέλο θα εκλεγεί μια χώρα. Οι πόλεις που συμμετάσχουν στον ανταγωνισμό αυτό τροποποιούνται. Καταβάλουν τεράστιες προσπάθειες. Προσπάθειες τι κάνουν βέβαια για να υποβάλουν την υποψηφιότητα, αλλά δεν είναι περιττές συνεχίζουν. Στη Γερμανία παραδείγματος χάρη είχαμε πολλές πόλεις που είχαν υποβάλει ψηφιότητα ταυτόχρονα με το ΕΣΕΝ. Οι πόλεις αυτές εξακολουθούν σήμερα να είναι ενωμένε μεταξύ τους. Δεν θέλω λοιπόν να παραμείνει ότι είναι περιττό. Όχι. Αυτές είναι προσπάθειες που δεν θα είχαν καταβληθεί και που γίνονται προς όφελος των πολιτών και προς όφελος των πόλεων. Μετά, έχω μια ερώτηση και συμφωνώ εδώ με την Έρικα Τρίπελ. Μέχρι το 2019 είναι όλα ε, κανονισμένα. Και το είχαμε ε, κάνει ήδη εκ αρχή. Εμείς το 1999 δεν ξέραμε ότι το 2004 θα είχαμε νέες χωρισμένοι και το 2007 άλλα δύο καινούρια και είχαμε πει μέχρι το 2019 μία στη χώρα, μία χώρα κάθε φορά. Και τελικά ε, αρχίσαμε και άρχισε το, το Λουξεμβούργο με μία χώρα από την Ανατολή της δύο δηλαδή. Επελέχθη από το Λουξεμβούργο. Εγώ αναρωτιέμαι τώρα τι θα γίνει μετά το 2019. Πιστεύετε ότι θα πρέπει να συνεχιστεί αυτή η μέθοδος. Μία πόλη κάθε χρόνο, δύο πόλεις κάθε χρόνο ή υπάρχουν και άλλες δυνατότητες. Ας πούμε, να πούμε μία περιοχή. Η κυρία Αντζικοσιόπ το έκανε αυτό με το Λουξεμβούργο. Ήταν δύσκολο. Το Μαστρίχ λέει τώρα ότι εάν συνενώσει όλη την περιοχή του θα μπορέσει να έχει μεγαλύτερο βάρος. Μέχρι το Άχεν. Αλλά αυτό δεν το λαμβάνει ιδιαίτερα υπόψη η Κομισιόν και θα μπορεί να μας πει και κάτι η Κομισιόν μετά. Τι θα γίνει μετά το 2019. Γιατί ε, αν έχουμε μία πόλη όπως ε, στο παρελθόν θα παράσουν δύο γενιές μέχρι να ξαναδοθεί η δυνατότητα σε μία χώρα. Δεν μπορεί να είναι αυτό το νόημα. Χάνεται αυτή η ιδιότητα της πόλης Φάρου. πρέπει να δούμε τι θα γίνει με το 2019. Να σκεφτούμε το θέμα της κριτικής επιτροπής. Όταν λέγεται ότι μπορεί κανένα να είναι τρία χρόνια μονάχα μέλο της κριτικής επιτροπής και μετά δεν μπορεί να παρακολουθήσει τι έγινε ή τι θα γίνει. Ήδη και αυτό δεν είναι καλό. Ίσως θα πρέπει να σκεφτούμε μήπω μπορούμε κάτι να αλλάξουμε. Αλλά έχω και μία, και μία ερώτηση. Η εποπτεία που γίνεται και που θέλαμε να υπάρχει είναι αποτελεσματική κατά τη γνώμη σας. Να δω. Να πάω σε μια χώρα που ήταν η τρίτη. Κωνσταντινούπολη είχε υποβάλει μια θαυμάσια πρόταση. Το θυμάμαι αυτό. Από ανθρώπους από τις μη κυβερνικέ οργανώσεις, από την κοινωνία των πολιτών κλπ. Και όταν έγινε πολιτιστική πρωτεύουσα δεν είχαν καθόλου λόγο. Μόνο κάποιες επιχειρήσεις, η ίδια η πόλη επιβλήθη... Αυτό δεν επιτρέπεται να γίνεται. Μπορείτε να το παρεμποδίσετε. Αρκεί η υποπτία. Πολλές ερωτήσεις βέβαια. Κάποιος άλλος που έχει να υποβάλει μια ερώτηση. Αλλιώς θα δώσω δυνατότητα στο πάνελ να απαντήσει. Κύριε Βίζαντ. Herr nein, αφού είχατε την ευγενή καλοσύνη να αφαιρθείτε σε μένα. Κοιτάξτε, εγώ δεν είμαι σε καμία περίπτωση κατά του ανταγωνισμού ή του συναγωνισμού, αλλά ε, εγώ το διατύπωσα και πάρα πολύ προσεκτικά στο κείμενό μου. Είναι η δεύτερη παύλα, ε, ε, στην πρώτη παράγραφο, στο α. Σε κάθε περίπτωση ήταν χρήσιμο. Και είναι τεράστια διαφορά από περίπτωση σε περίπτωση. Εγώ σας έφερα την πολιτισμόν στο Βέλγιο και το Κόζιτσε στη Μόνς αν αναλάβει πολιτιστική πρωτεύουσα το 2015 θα έχει μέχρι τότε μία δεκαετία περίπου για να τα προετοιμάσει όλα σωστά. Γιατί ήξερε από πολύ νωρί ότι θα υποστηριχθεί, ότι θα είναι πολιτιστική πρωτεύουσα το 2015 και δεν υπήρχε ανταγωνισμός. Αυτό είναι κρίμα όμως. Και γι' αυτό δεν υπερψήφισα ε, ε, παρόδο, το λέω αυτό, στον πρώτο γύρο, την πρόταση αυτή, αλλά όταν πήγαμε επί τόπου ε, και είδαμε ποια επιτυχία είχε και με την παρακολούθηση επίστην. Δηλαδή, η καλή προετοιμασία πραγματικά έχει νόημα. Ίσως θα μπορούσαμε έτσι να το αναφέρουμε, να συμφωνήσουμε σε αυτό ότι χρειάζεται περισσότερη προετοιμασία αλλά και δεσμευτική κατά κάποιο τρόπο. Το είπα και προηγουμένως. όταν κάποιος δεσμεύεται θα πρέπει να υλοποιεί και αυτά για τα οποία έχει δεσμευτεί. Αυτό είναι πολύ σημαντικό στην όλη αυτή η ιστορία. Μπορούμε λοιπόν να το παρακολουθήσουμε, προσπαθήσαμε στην παρακολούθηση να το κάνουμε, στο monitoring όπως λέγεται, και οι διάφορες ε, διαδικασίες και επιλογές έχουν αλλάξει και αλλάζουν συνεχώς για να προσαρμόζονται. Δεχτήκαμε και τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αναφέρθηκε αυτό προηγουμένως, αλλά είναι πραγματικά πολύ μικρή η μονάδα. Το τμήμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που φορτίζεται με αυτό το έργο είναι πολύ μικρή υπηρεσία. Γιατί δεν είναι δύο, τρεις ή τέσσερις υποψηφιότητες, αλλά ξαφνικά πολλαπλασιάζονται, όπως στην περίπτωση της Πολωνίας και της Ισπανίας και υφίστανται και οι ίδιοι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τεράστια πίαση, όπως και εμείς στην ε, Κριτική Επιτροπή. Αυτό κάπου θα πρέπει να βρίσκεται ανάκλαση στους μελλοντικούς κανόνες με ε, προσαρμογή κάποιων θεμάτων και πιο μεγάλη ευελιξία. Η κυρία Πακ. Για την περίοδο μετά το 2019 δεν έχετε πρόταση. Η κυρία Γλάντης. To ε, αναφερθήκατε στο έγγραφο το οποίο είναι πολύ ευρύτερο από τα συμπεράσματα γιατί αφορά και κάποιες σκέψεις για την ευρωπαϊκή πολιτική. Μάλιστα. 2,8 εκατομμύρια ήταν οι απασχολούμενοι το 2006 στον πολιτισμό. Καταλαβαίνετε ότι είναι μεγάλο κλάδος της οικονομίας. Και επίσης, επειδή η παραδοσιακή οικονομία γνωρίζει κρίση τώρα, ίσως η κινητήρια δύναμη της ανάπτυξης να είναι ο πολιτισμός τώρα. Αυτά που σας λέω μπορεί να είναι κοινότυπα. Ε, αλλά τα γνωρίζουμε όλοι. Ας πούμε, η Κρακοβία όταν έγινε το 2000 πολιτιστική πρωτεύουσα είχε 1,3 εκατομμύρια ε, ε, επισκέπτες το χρόνο. Ε, μετά τον επόμενο χρόνο αυτοί έγιναν 1,4 εκατομμύρια και συνεχώς αυξανόταν ο αριθμός των επισκεπτών και έχουν φτάσει φέτος στα 7-8 εκατομμύρια. Πραγματικά χρειάζεται επενδύσεις ο πολιτισμό και ενίσχυση και σιγά σιγά προχωρήσει. σε ό,τι αφορά το λεγόμενο Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Μήνα, έχω απογοητευτεί πάρα πολύ και ζητώ συγγνώμη που το λέω εδώ. Ήταν πολύ καλή πρωτοβουλία αυτή, ευρωπαϊκή, αλλά σταμάτησε κάποια στιγμή και δεν ανανεώθηκε, δεν αναζωογονήθηκε. Εμείς ως Ευρώπη θα πρέπει κανονικά να έχουμε ένα πρόγραμμα που να απευθύνεται στις γειτονικές μας χώρες, χώρες που προσδοκούν να γίνουν μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διευκολύνει και την κατανόηση και το δημοκρατικό μετασχηματισμό. Και μπορώ να σας τα πω αυτά εγώ ως Πολωνή. Έχω ζήσει ακριβώς το ίδιο στο πετσί μου, για να το πω έτσι. Ίσως τα επόμενα χρόνια να δοθεί νέα πνοή σε αυτό τον Ευρωπαϊκό, Ευρωπαϊκό, Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Μήνα όπου να συμμετέχουν χώρες και από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και εκτός της Ένωσης. Χρειαζόμαστε αυτό το διάλογο των πολιτισμών και τη συνεργασία με άλλους. Γι' αυτό στα συμπεράσματά μου θα ήθελα να φέρω και το αναφέρω άλλωστε αυτό, να επαναφέρουμε τον ε, Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Μήνα. Α, ξέχασα να απαντήσω σε αυτό το θέμα των πολιτικών ή πολιτιστικών κριτηρίων που ετέθη προηγουμένως. Σε κάποιες χώρες, όπου αυτό ήταν ένα ζήτημα, από ό,τι φαίνεται, είχαμε εσωτερικέ συζητήσεις και είχαμε πάρει μια απόφαση ε, πολύ σοβαρή και πολύ αυστηρή. Όποτε το θέμα γινόταν πολιτικό και η συζήτηση γινούσε στα πολιτικά, τη διακόπταμε και ε, επιστρέφαμε στα πολιτιστικά κριτήρια για την επιλογή της πολιτιστικής πρωτεύουσας. Νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό Για να το τονίσουμε ως απάντηση στην προηγούμενη ερώτηση που Βεβαίως και δεν είμαστε υπεύθυνοι για το ότι λέγουν κάποιοι εκτός, ότι τύπος, πώς προβάλλεται αυτό οι πρωτεύουσε, οι πόλει μπορεί να το προβάλλουν όπω θέλουν. Αυτό είναι άλλη υπόθεση. Ούτε εμεί είμαστε υπόλογοι. Εάν, για παράδειγμα, βγει ένα υπουργό και πει ότι θα πρέπει να γίνει πολιτιστική πρωτεύουσα η Α ή Β πόλη, δημοσίω, πριν εμεί αποφασίσουμε. Δεν είναι δική μα υπόθεση αυτό, ούτε δικό μα φταίξιμο. Αλλά προσπαθούμε να αποφεύγουμε αυτέ τι πολιτικέ συζητήσει μέσα στο πάνελ. Και μια που με ρωτήσατε για το διάστημα μετά το 19, πιστεύω ότι πραγματικά οι πολιτιστικές δραστηριότητες θα πρέπει να καλύπτουν όλη την Ευρώπη, γιατί είναι και κοινή η ιστορία μας άλλωστε. Αλλά αμφιβάλλω κατά πόσο γίνεται αυτό στο παρόν σύστημα. Ευχαριστώ. Θεωρώ der Länderturnus keine schlechte Sache war. ότι αυτές οι δύο πόλεις από την παλιά και την νέα Ευρώπη αν θέλουμε να το πούμε έτσι που επιλέγονται ταυτόχρονα είναι καλό γιατί υπάρχει μια στενή συνεργασία μεταξύ αυτών των δύο εκλεγμένων πόλεων. Αυτό ήταν ένα τμήμα του προγράμματος. Όσον αφορά τώρα την εποπτεία. Η Κριτική Επιτροπή έπαιξε πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Είχαμε πει σε διευθυντές, υπέστητος για την πολιτιστική ε, πρωτεύουσα ότι εάν κάποια στιγμή δεν κάνετε έκκληση στην ε, δεν μπορούσαν να κάνουν έκκληση να έρθουν σε επαφή με την κριτική επιτροπή θα είχε αποτύχει όλη η διαδικασία αλλά πρέπει να δούμε ποια είναι η θέση αυτής της κριτικής επιτροπής ε, το κάνουμε εμείς έτσι παράλληλα με τις άλλες εργασίες μας. Αλλά θα πρέπει να δούμε ότι αυτό το σώμα, αν δεν είναι πια διαγωνισμός, δεν χρειάζεται να το λέμε κριτική επιτροπή, αλλά αυτό το σώμα θα πρέπει στο μέλλον να έχει ίσως άλλη μορφή. Θεωρώ ότι θα πρέπει να παίξουν σημαντικότερο ρόλο οι χώρες, γιατί θα πρέπει τα εθνικά κράτη να αναλάβουν τις ευθύνες τους. η πολιτική ε, διαμάχη, δηλαδή κομματική πολιτική εννοούμε, πολιτική είναι το πιο ευγενικό τμήμα, θέλετε, και όταν έχουμε ε, πραγματική ευγενή πολιτική, δεν μπορούμε να ξεχάσουμε τον πολιτισμό. Απ' την άλλη μεριά, εδώ είχαμε διαφορετικού τύπου πολιτική, δηλαδή ορίστηκε μια πόλη, έγιναν μεταξύ εκλογές, ανέλαβε κάποιο άλλο κόμμα την ε, ισχύ και υπήρχαν διαφορετικά προβλήματα ξαφνικά. Θα πρέπει εκεί λοιπόν να ε, δράσουμε καθησυχαστικά. Αυτό που κατηγορούν οι πόλεις κυρίως είναι η δυνατότητα πρόσβασης στις εμπειρίες των προηγουμένων πολιτιστικών πρωτευουσών. Και αυτό δεν πρέπει να το παραβλέπουμε, γιατί ένα δίκτυο μεταξύ των πολιτιστικών αυτών πρωτευουσών θα ήταν μια τεράστια πηγή ιδεών, πρωτοβουλειών και δυνατοτήτων. Λοιπόν, η διεύρυνση αποφασίστηκε το 2000, ε, ε Το 99 απλώς οι υπουργοί πήραν λάθος απόφαση. Ήταν γνωστό. Ε, για να ρωτήσω. Από όσο ξέρω, υπάρχει έντονη ανταλλαγή απόψε μεταξύ των παλιών πρωτεύουσων και των νέων που υποβάλλουν υποψηφιότητα. Το Μαστρίχ, παραδείγματο χάρη, που τώρα είναι η υποψήφια, ξέρω ότι πήγαν οι υπεύθυνοι στο Έσεν, στην Ιταλία, στο Τουρκού για να πάρουν τις διάφορες εμπειρίες. Ναι, αυτό είναι ένα ανεπίσημο, ανεπίσημο λέω δίκτυο. Αν ήταν όμως δομημένο, να υπάρχει δηλαδή κάποιο βήμα, κάτι οργανωμένο για να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων, θα ήταν καλύτερο. Γίνεται, γίνεται, όπως είπες, αλλά αυτό είναι η δύο πρωτοβουλία. Πρόεδρος, εντάξει, αυτό είναι μια πρόταση προς την Κομισιό να το κάνει αυτό στο μέλλον. Στον έχει το λόγο. Εγώ ήθελα να ρωτήσω, γιατί δεν κατάλαβα καλά μια διαδικασία. Αυτό που ζήτησε και ο συνάδελφος Σαντιάγκο δηλαδή, αλλά δεν το απάντησαν. Στις σημειώσεις που μας μοιράστηκαν από το 2013, διαδικασία που θα ξεκινήσει το 2013 μέχρι το 2019, το κράτος μέλος ορίζει de facto μία πόλη. Δηλαδή, να καταλάβω καλά, ο ρόλος που είχαμε εμείς ως Κοινοβούλιο και ως Ευρωπαϊκή Ένωση και το Συμβούλιο και η Κομισιόν δεν κάνουμε τίποτα άλλο παρά απλώς να καταγράφουμε αυτό που αποφασίζει το κράτος μέλος. θα έπρεπε ίσως αν δεν μπορούμε να αλλάξουμε αυτή τη διαδικασία από το 2019 και μετά να φανταστούμε έναν πιο δυναμικό ρόλο των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων όπως είχε γίνει και παλιότερα ούτως ώστε να έρχονται από το κράτος μέλος τουλάχιστον δύο προτάσεις και μετά το πάνελ των εμπειρογνώμων θα αποφασίσει ποια από τις πόλεις είναι η καλύτερη και αυτό ανάλογα και με τις δικές μας σκοπιμότητες ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Μου φάνηκε ενδιαφέρουσα η πρόταση της συναδέλφου να φανταστούμε ότι θα μπορούσαμε κάπου αυτό το σκεπτικό να το διευρύνουμε. Εγώ αυτούς τους μήνες διαπιστώνω ότι ορισμένες υποψηφιότητες για το μέλλον προβλέπουν μία... Όχι μόνο ένα άνοιγμα της ίδιας της πόλης που προτείνεται, αλλά ε, ένα άνοιγμα ευρύτερο, περιφερειακό, ε, με άλλες ε, ή μέσα από άλλες πόλεις, κοντινές πόλεις θα μπορούσαμε να έχουμε δηλαδή μια τέτοια διάσταση από το 2019 και μετά. Μάλιστα. Σήμερα το πρωί κάναμε αυτό που επιτρέπεται κύριε Φίσα που ρωτήσατε. Δηλαδή αυτό που κάναμε σήμερα το πρωί ήταν η αρμοδιότητά μα. Δεχτήκαμε την πρόταση για το Βρότσλαφ και το Σαν Σεμπαστιάν. Είναι η πρόταση. Εμείς δεν είμαστε ειδικοί εμπειρογνώμονες, παρακολουθούμε, ελέγχουμε, δεν κρίνουμε. Είναι διαδικαστικό αυτό, έτσι, και τίποτα παραπάνω. Αλλά θα πρέπει να γίνει, διότι είναι μια κοινή δράση μας. Για μένα είναι λίγο προβληματικό αυτό. Δεν ξέρω γιατί το πίστεψα, αλλά ανέκαθεν θεωρούσα ότι κάθε χώρα θα πρέπει να προτείνει τουλάχιστον δύο πόλεις, δύο υποψηφιότητες, για να υπάρξει επιλογή. Δεν ξέρω, λάθος το κατάλαβα. Μήπως δεν κατάλαβα σωστά αυτά που έχετε γράψει εδώ. Γιατί είναι τρελό. Η Κριτική Επιτροπή μπορεί να επιλέξει, αλλά αν είναι μία πρόταση μόνο, θα πει ότι δεν μας κάνει αυτή η πρόταση. Και τι θα γίνει. Θυμάστε με την Πάτρα τι είχε γίνει. Ήταν τρελό. Ο κύριος Ροκάρο, προκάτοχός μου, είχε βγει από τα ρούχα του. Γιατί δεν κατάλαβε γιατί η Ελλάδα είχε προτείνει την Πάτρα για πολιτιστική πρωτεύουσα και προσπαθούσε να πείσει τους ε, δικούς του στο κόμμα του και στην Πάτρα που ήταν για αυτοί εκεί πέρα σοσιαλιστές να το αποσύρουν. Δεν υπήρχε άλλη πρόταση. Και εμείς θέλουμε να έχουμε δύο ε, προτάσεις από κάθε χώρα. Για να ξανάρθουμε στη Γερμανία είχαμε μια τεράστια λίστα υποψηφίων, δεν θυμάμαι 8, 10 και παραπάνω, που ήθελαν να είναι πολιτιστική πρωτεύουσα και η Γερμανία επέλεξε. Πώς το λέγανε αυτό και το γερμανοπολωνικό. Πώς το λένε. Γκέρλιτς. Μπράβο. Και, και την πόλη του Έσεν δεν επέλεξε. Η Γερμανία έκανε πρόταση δύο πόλεων και επέλεξε κριτική επιτροπή. Που ήταν αρκετά δύσκολο να γίνει επιλογή από δύο για τη Γερμανία. Για να επιλέξετε εσείς τελικά. Δεν ξέρω τι γίνεται. Θα μπορούσε κάποιος να μας διαφωτίσει ίσως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ας μιλήσει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μπορεί να μας ε, δώσει και καμιά ιδέα για το τι σκέφτεται για το μέλλον. Ο Σούχα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Τι να σας πω εγώ τώρα, να απαντήσω για αυτό το συγκεκριμένο ή γενικά. Για αυτό το συγκεκριμένο. Τώρα βρισκόμαστε σε ένα σύστημα το οποίο έχει ιδρυθεί μετά από απόφαση Κοινοβουλίου και Συμβουλίου το 2006. Είναι γεγονός ότι τα κράτη-μέλη από το 2013 και μετά είναι η Γαλλία και η Σλοβακία. Το Κόζιτσε και η Μασαλία ταυτόχρονα. Αλλά η επιλογή έχει αρχίσει ήδη από το 2007 με αυτό το νέο σύστημα ή τους νέους κανόνες. Ήταν οι δύο πρώτες χώρες. Και τώρα έχουμε υποχρεωτικό διαγωνισμό σε κάθε χώρα. Και είναι ένα διαγωνισμό, όπως ορίζει η απόφαση, από τη βάση προς την κορυφή. Δηλαδή, δεν κατεβαίνει μια χώρα με μια πρόταση. Είναι υποχρεωμένη η χώρα να κάνει διαγωνισμό, ε, να ανοίξει, να το προκυρήσει έξι χρόνια πριν για υποβολή υποψηφιωτήτων με μια φάση προεπιλογη και ορίζεται σαφώ ότι είναι ένα συνδυασμός εθνικών και ευρωπαϊκών μάλλον εμπειρογνωμών και τελικά ε, το επόμενο χρόνο γίνεται η επιλογή. Πάντα λοιπόν εφαρμόζεται αυτό από το 2007 μέχρι το 2013 και μετά. Μάλλον από το 2013 και μετά. Αναφερθήκατε στην περίπτωση του ΠΕΤΣ και του ΕΣΕΝ αυτό ήταν η προηγούμενη επιλογή. Ε, με άλλη μορφή, εθελοντικά τα κράτη είτε έκαναν επιλογές και διαγωνισμούς όπως έκανε η Γερμανία έκαναν ε, δύο προτάσεις τελικές, αλλά τον ίδιο χρόνο ήρθε το ΠΕΤΣ ως μοναδική υποψηφιότητα, οπότε τι να αποφασίσει η Κριτική Επιτροπή. Γι' αυτό λοιπόν κατέληξαν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στον υποχρεωτικό διαγωνισμό και από το 7 και μετά είχαμε μόνο μία περίπτωση ε, που ήταν μοναδική υποψηφιότητα και αυτή ήταν η περίπτωση του Βελγίου. Και σε αυτή όμως την περίπτωση ε, προκηρύχθηκε διαγωνισμός, αλλά κατατέθηκε μία και μόνη υποψηφιότητα. Και είχαμε αυτές τις δύο φάσεις προεπιλογής και επιλογής. Ήταν η μόνη περίπτωση από το 2007 και δεύτερον. Αλλά από τότε έχουμε τουλάχιστον δύο υποψηφιότητες και η περίπτωση της Ισπανίας είναι ακραία με 16 υποψηφιότητε. Αλλά τώρα η περίοδος αυτή ε, διαρκεί μέχρι το 2019 με το νέο σύστημα και τους κανόνες του 2006 και τη σχετική απόφαση. Η απόφαση του 2006 ορίζει ότι κάθε χώρα πρέπει να κάνει τουλάχιστον δύο προτάσεις. Σωστά το κατάλαβα. Όχι. Α, ούτε καν αυτό. Ε, μα καλά λάθος, θα καταλαβαίνω. Λοιπόν, κοιτάξτε, η απόφαση του 2006 ορίζει ότι ο διαγωνισμό θα πρέπει να γίνεται στο ιστορικό των κρατών μελών από κάτω προ τα πάνω, Χωρί καμία απέτηση για το ελάχιστο. Δηλαδή είναι από τη βάση προ την κορυφή, αν δεν υποβληθούν τουλάχιστον δύο υποψηφιότητε, δεν θα του το επιβάλλετε. Όσοι καταθέσουν υποψηφιότητα, Σα είπα στο Βέλγιο κατατέθηκε μόνο μία. Σε όλες τις υπόλοιπες χώρες ήταν τουλάχιστον δύο, στη ΔΕ Ισπανία 16. Ναι, αλλά κύριε Σούχαρ μου. Γνώμη που επανέρχομαι. Θα γίνει διαγωνισμό στο εσωτερικό των κρατών μέλων. Μπορεί, δίνανται, οφείλουν, ξέρω εγώ, εντάξει. Τελικά, η χώρα, αν έχει τη δυνατότητα, αν υπάρχει μία και μόνη υποψηφιότητα, είναι ανόητο. Ωραία. Ε, ε, η χώρα είναι υποχρεωμένη να καταθέσει τουλάχιστον δύο ε, προτάσεις στην Κριτική Επιτροπή. Μπορεί να είναι και μία αυτή. Όχι. Οι χώρε δεν υποβάλλουν πρόταση στην κριτική Επιτροπή. Οι προτάσει υποβάλλονται στην ενωμένη αυτή κριτική επιτροπή, ευρωπαϊκή και εθνική. Είναι μια κοινή δηλαδή συνάντηση της Κριτικής επιτροπή του κράτου και της Ευρώπης και γίνεται εκεί η προεπιλογή και μετά υποβάλλεται επίσημα η πρόταση στην κυβέρνηση του κράτους μέλους. Η κυβέρνηση του κράτους μέλους έχει την υποχρέωση να προτείνει μία πόλη στο Συμβούλιο. Και ο ρόλος του Κοινοβουλίου είναι ότι το Κοινοβούλιο έχει το δικαίωμα να ορίσει δύο μέλη στην Ευρωπαϊκή Κριτική Επιτροπή και γνωμοδοτεί το Κοινοβούλιο για τις επιλογές αυτές. Αυτή είναι η κανόνας. Πρόεδρος, πάλι δεν τα κατάλαβα. Οι άλλοι ίσως τα κατάλαβαν, εγώ δεν κατάλαβα τίποτα, θα μου το εξηγήσουν κατευθείαν. Α, και ο κύριος Φίσης δεν κατάλαβε. Για να το εξηγήσω στα, στα γερμανικά ίσως. Έγινε μια αλλαγή διαδικασίας μεταξύ της επιλογής όπως είχε γίνει τότε στη Γερμανία με μια προκαταρτική επιλογή στο εσωτερικό της χώρας που κατέληξε στους υποψηφίους. Σήμερα δεν υπάρχει αυτό το φιλτράρισμα. Γι' αυτό είναι δυνατόν οι 16 που είχαμε στη Γερμανία τότε μπορούν άμεσα να υποβάλουν υποψηφιότητα. Αυτή είναι η διαφορά. Και μετά υπάρχει αυτή η φάση της προεπιλογής που από τις 16 καταλήγουν σε 4, 5 ή 2 που μπορούν να προωθήσουν επίσημα την υποψηφιότητά τους. Η, η βάση μας θα διαφορετική. Σαντιάκο το κατάλαβες κι εσύ. Άλλοι ξανά. Όλοι μπορούμε. Μπορούν να υποβάλουν την υποψηφιότητα από την ελόγω χώρα και η Κριτική Επιτροπή έχει το έργο από τι 16, 17, 20 χώρε να επιλέξει, ε, πόλεις να επιλέξει μία. Η χώρα δηλαδή έχει το δικαίωμα να αποκτήσει την πρωτεύουσα αυτή την πολιτιστική. Αλλά οι πόλεις, οι πόλεις υποβάλλουν την ψηφιότητα σε εσά. Εντάξει, ωραία. So, äh, möchte die Kommission äh, weitergehende Ausführungen zu nach 2019 machen. Λοιπόν, τι θα γίνει τώρα μετά το 2019. Ποιος θα απαντήσει από την Κομισιόν. Okay, thank you. Thank you, Madam Chair. I'm not, uh, I don't think that I'm going to Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν νομίζω ότι θα σας διαφωτίσω για το τι θα γίνει με το 2019. Γιατί δεν υπάρχει απόφαση της Κομισιόν. Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ποια είναι η διαδικασία, τι κάνουμε. Εκτιμώ βέβαια τη δική σας πρωτοβουλία να οργανώσετε αυτή την ακρόαση. γιατί είναι ένα άλλο πετραδάκι στο μοσαϊκό που εξετάζουμε. Έχουμε διαβουλεύσεις online με συμμετοχή έντονη, έχουμε δημοσιεύσει τα αποτελέσματα, είχαμε μια δημόσια ακρόαση στις Βρυξέλλες ε, το Μάρτι. Έχουμε τις εκθέσεις αξιολόγησης ε, για τις ε, τώρα οι μετά την δηλαδή, του 2006 υπάρχουν διάφορες ε, πηγές που λαμβάνουν υπόψη κατά τη διάρκεια δημιουργίας μιας άποψη και μιας προετοιμασία απόφαση. Έχουμε 7 μέλη στο πάνελ και είμαστε σε συνεχή επαφή μαζί του, και το θέμα της επόμενη χρονικής περίοδου ε, εξετάζεται συνεχώς. Θα ήθελα, Πρόεδρε, να επανέλθω στην ερώτησή σας, γιατί κανένας δεν απάντησε για το θέμα της εποπτείας. Ρωτήστε κατά πόσο η εποπτεία που αναφέρεται στην απόφαση του 2006 λειτουργεί σωστά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο και η εισαγωγή της υποχρέωσης ε, εποπτείας ε, στην απόφαση ήταν πάρα πολύ σημαντική. Και η απόφαση αυτή κατόπιν ε, ε, πρόταση του πάνελ ε, διευρύθηκε με μια ανεπίσημη αποπτία, όπως τη λέμε. Έχουμε μια πρώτη φάση δηλαδή εποπτείας ε, που είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο και θα είναι και στη μελλοντική πρόταση της Κομισιόν. Η ανεξαρτησία της Επιτροπής είναι πάρα πολύ σημαντική και σίγουρα θα προτείνουμε ένα ευρωπαϊκό πάνελ και μια ευρωπαϊκή κριτική επιτροπή γιατί υπήρχε πάντα εκεί υψηλού επίπεδου καλλιτεχνική ε, πραγματογνωμοσύνη αλλά και ανεξαρτησία και ουδετερότητα. Και εκεί βρίσκεται νομίζω ο κρόγωνιος λήθος για την επιτυχία του ευρωπαϊκού πάνελ. που έτσι εγγυάται τις επιλογές που έχουν γίνει μέχρι στιγμές. Και αυτό είναι κάτι που θα συμπληρευτεί επίσης στην μελλοντική πρόταση. Η δικτύωση αναφέρθηκε σε ένα σημαντικό στοιχείο για το μέλλον. Ναι, πράγματι, έχετε δίκιο. Υπάρχει ένα δίκτυο πόλεων, είναι ανεπίσημο το δίκτυο αυτή τη στιγμή και τις έχουμε καλέσει πολλές φορές. Ε, ε, το 2007 πρώτη φορά νομίζω τους καλέσαμε σαν κομισιόν, ως κομισιόν και τους είπαμε θέλετε να κάνουμε εμεί κάποιες ειδικέ προσκλήσεις για να επισημοποιήσετε το δίκτυο σας. Πάντα μας είπαν όχι, όχι, δεν θέλουμε να έχουμε καμία επισημοποίηση. Θέλουμε να παραμείνει ανεπίσημο το δίκτυο αυτό. Και το δίκτυο ε, προεδρεύεται από την πόλη στην οποία συνεδριάζουν. Και δεν θέλουν να έχει οπωσδήποτε παρουσία η Επιτροπή εκεί, γιατί αναφέρουν τις επιτυχίες τους αλλά και τις αποτυχίες τους, τα προβλήματα και γι' αυτό δεν θέλουμε να παρέμβουμε, γιατί βλέπουμε ότι μέχρι στιγμή λειτουργεί πολύ θετικά. Όσον αφορά την ευρωπαϊκή διάσταση, βέβαια στην απόφαση υπάρχει μία παράγραφος για την ευρωπαϊκή διάσταση και μπορώ κάλλιστα να συμφωνήσω με όλα τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής που έφτιαξαν το θέμα αυτό. Από την άλλη μεριά είναι πάρα πολύ δύσκολο να είμαστε πιο συγκεκριμένοι γιατί έχουμε μεγάλη ε, διαφοροποίηση στην Ευρώπη. Έχουμε μεγάλες χώρες μεγάλες πόλεις, έχουμε μικρές πόλεις και έχουμε μικροσκοπικές πόλεις που υποβάλλουν ε, υποψηφιότητα. Έχουμε πόλεις στο κέντρο, έχουμε πόλεις στην περιφέρεια. Η ευρωπαϊκή δράση λοιπόν είναι πάρα πολύ διαφοροποιημένη. Δηλαδή η ευρωπαϊκή διάθεση στο Ταλίν είναι πολύ διαφορετική από την ευρωπαϊκή διάθεση στη Μασαλία. Και εάν εμείς ορίσουμε δείκτες ή κάποια άλλα στοιχεία για να ποσοποιήσουμε αυτή την ε, ευρωπαϊκή διάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολο. Θα πρέπει λοιπόν να υπερβάλλουμε γιατί είναι όπως σας είπα πάρα πολύ διαφοροποιημένο στοιχείο αυτή η ευρωπαϊκή διάσταση και δεν αφορά μόνο τον αριθμό των αλλοδαπών που υπάρχουν σε αυτή την πόλη. Υπάρχει και το θέμα της οικονομικής επίπτωσης ε, τη ιδιότητας ε, πολιτιστική πρωτεύουσα. Είχαμε μια σειρά μελετών που είχαν συγκεντρωθεί σε αυτό, η πρώτη το 2005, που το αφορούσε τις πολιτιστικές πρωτεύουσες και μόνο. Το 2006 είχαμε μια μελέτη για την οικονομία της, ε, του πολιτισμού που συμμετείχαν και οι πρωτεύουσες και ε, μετά είχαμε και μια μελέτη για την δημιουργικότητα όπου χρησιμοποίησαμε στοιχεία από διάφορε πολιτιστικέ ε, πρωτεύουσε και είχαμε την υποχρεωτική εξωτερική αξιολόγηση των πόλεων κάθε χρόνο και την ε, οικονομική επίπτωση την αξιολογούμε κάθε φορά. Νομίζω λοιπόν ότι οι ευρωπαϊκέ πολιτικέ ε, πρωτεύουσε είναι οι δραστηριότητε τη Ευρωπαϊκή Ένωση, την οποία έχουν περισσότερα στοιχεία για τι οικονομικέ επιπτώσει. Πρόεδρο, Έχω και μια ερώτηση. Αναφερθήκα σε μια Ευρωπαϊκή Κριτική Επιτροπή. Ε, τι άλλο δηλαδή. Είπατε πρέπει να έχουμε μια Ευρωπαϊκή Κριτική Επιτροπή. Δεν κατάλαβα, δεν άκουσα ποτέ να θέλει κανένα να προσκαλέσει Αμερικανού ή Ασιάτε. Ή σα παρεξήγησα κάπου. Τι εννοούσατε όταν αναφερθήκατε στην Ευρωπαϊκή Κριτική Επιτροπή. Okay. Μάλιστα, να σας πω. Τώρα έχουμε δύο είδους κριτικές επιτροπές που συνεργάζονται. Η μία είναι ευρωπαϊκή, που διορίζεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Επιτροπή Περιφέρειων και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και μετά έχουμε και την Εθνική Κριτική Επιτροπή. Αυτό που σα ανέφερα ήταν ακριβώ η Ευρωπαϊκή, που εδώ ε, ε, έχετε ενώπιον σα τρει εκπροσώπου τη, οι οποίοι είναι πιο σημαντική ε, και διασφαλίζει την ακαιρεότητα και τη δικαιοσύνη του συστήματος. Α, εγώ το είχα αντιληφθεί αλλιώ στο ευρωπαϊκό, όχι οι Αμερικανοί ή οι Ασιάτες. Ε, όχι, δεν προτείνουμε ακόμα να φέρουμε Αμερικανούς για την Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Πρωτεύουσα. Ναι, ο κύριος Βίζαντ, ε, θα ήθελα μια που τόνισε το ρόλο της Κριτικής Επιτροπής η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν θα ήταν ε, κακό να πάω αυτή τη μικρή πρόταση. Το πάνελ να μην είναι μόνο Βρετανή και Αυστριακή. Έγινε μια ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των διαφόρων ε, οργανισμών. Καλό είναι να εκπροσωπείται ολόκληρη η Ευρώπη. Η πρόεδρος, ε, μα το Κοινοβούλιο πιστεύω καταβάλει πάντα προσπάθειες. Ε, δεν μπορούμε να καλύψουμε με αυτούς τους δύο τους πάντες. Ίσως να το πούμε και στις κυβερνήσεις και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να είναι μεγαλύτερο το φάσμα γιατί η ευρωπαϊκή πολιτιστική διάσταση ορίζεται τουλάχιστον από τους 27 συν τους άλλους που θέλουν να προσχωρήσουν. Σας ευχαριστώ πολύ που ε, το επισημάνατε, που δείξατε ότι αυτό το δίκτυο συνεδριάζει τρεις ετησίως σε διάφορα μέρη. Είναι ένα χαλαρό δίκτυο. Καλό είναι να μην δεσμευτεί κανείς έτσι πάρα πολύ άκαμπτα. Η ιδέα αυτή της εθελούσιας συμμετοχής να παραμείνει και να διαφυλαχθεί. Καλό είναι αυτό. Λοιπόν, παραμένει ακόμα μία ερώτηση. Δεν, δεν μου απαντάει κανείς σήμερα. Τι είναι αυτό το πρόβλημα. Μετά το 2019 πώς θα έχει η κατάσταση. Θα είμαστε σε θέση. Να το πω αλλιώς. Μετά το 2009 έχω την αίσθηση ότι δεν μπορούμε να επιστρέψουμε στο παρελθόν και να πούμε μία και μόνη πολιτιστική πρωτεύουσα, γιατί ο καθένας θα έχει σειρά μετά από 27 χρόνια. Ε, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Έχουμε καμιά ιδέα τι θέλουμε. Δύο χώρες το χρόνο. Ξανά. Ή αυτές οι χώρες που είναι σε μια ευρωπαϊκή πορεία, ανεξάρτητα από το που βρίσκονται προεταξιακά, παράδειγμα τα Δυτικά Βαλκάνια. Να έχουν την ευκαιρία και αυτοί να υποβάλουν υποψηφιότητα ή δεν μας έχει προβληματίσει. Δεν χρειάζεται να δεσμευτείτε, αλλά να το σκεφτείτε, σας ζητώ. Βεβαίως, κυρία Πρόεδρε, είναι όλες αυτές οι επιλογές που εξετάζουμε και αξιολογούμε και σίγουρα δεν πρόκειται να προτείνουμε μία απόλυτο χρόνο, τουλάχιστον δύο, όπως έχει τώρα η κατάσταση, ίσως και περισσότερες αξιολογούμε, ε, μελετούμε, δοκιμάζουμε διάφορες δυνατότητες, εκπεριτροπή συστήματα, ομάδες κρατών. Όλα αυτά είναι τμήμα της μελέτης αντικτύπου που θα δημοσιευθεί ως έγγραφο ιστορικό εργασίας Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Για να δείτε ποια είναι η σκέψη μας, η αξιολόγηση, ο προβληματισμός, θα κάνουμε όσο γίνεται καλύτερη πρόταση. Βεβαίω, λαμβάνουμε υπόψη και το μεγάλο ενδιαφέρον και ότι η ευρωπαϊκή πολιτιστική διάσταση δεν αφορά μόνο τα 27 κράτη-μέλη και ο ευρωπαϊκός πολιτισμός. Ε, μας προβληματίζει αυτό και σκεφτόμαστε πώ μπορούμε αυτή τη διεθνή διάσταση των υποψηφίων χωρών και των υπολείπων να τη λάβουμε υπόψη μας. Επίσης, ε, σε μια διαβούλευση που έγινε στο διαδίκτυο, εκδηλώθηκε μεγάλο ενδιαφέρον για τη συμμετοχή και των τρίτων χωρών και σίγουρα δεν πρόκειται να το αγνοήσετε. Ωραία, είστε τότε σε καλό δρόμο, λέει η Πρόεδρο. Άλλη ερώτηση, ο Σαντιάγκο. Εγώ ίσω πια να γίνομαι λίγο βαρύ. Γιατί ε, έχω κατά νου του θέματα με το... Με τον αθλη... με απασχόλησαν θέματα με τον αθλητισμό. Είχα και ακροασει Τώρα εγώ δεν μπορώ όμως να πω ναι σε κάτι που με προτείνουν χωρίς να μου το εξηγήσουν. Δηλαδή τι κάνουν, μας προτείνουν εδώ μια υποψηφιότητα και άντε εμείς τη δεχόμαστε σε αυτήν την επιτροπή. Μα αυτό δεν, δεν, δεν, δεν είναι εκλογή, επικύρωση είναι και άμα δεν μ' αρέσει τι κάνω. Δηλαδή δεν μπορώ να πω όχι γιατί δεν έχω και άλλη επιλογή. Δεν ξέρω μήπως θα έπρεπε δηλαδή να, να, να προτείνει ένα κράτος μέλος δύο πόλεις και άμα δεν έχει τότε έξω. Ας έρθει άλλη χώρα να μας προτείνει δύο. Αλλά έτσι μας αρέσει, δεν μας αρέσει, χωρίς καμία εξήγηση στα καλά του καθουμένου, δεν μου φαίνεται ένα σωστό σύστημα. Λοιπόν, θα πρέπει να δούμε. Κάθε χώρα που επιλέγεται έχει το δικαίωμα να αποκτήσει μία χώρα ως πολιτιστική πρωτεύουσα. Τώρα, οι πόλεις που θέλουν να γίνουν πολιτιστικές πρωτεύουσες πρέπει να υποβάλουν υποψηφιότητα. Όχι στη Μαδρίτη, στην πρωτεύουσα τους, ας πούμε, αλλά στην Κομισιόν και στην ε, Κριτική Επιτροπή. Η Κριτική Επιτροπή κάνει την επιλογή. Εμείς συμμετέχουμε, όπως και το Συμβούλιο, γιατί αποστέλουμε εμπειρογνώμονες στη κριτική αυτή επιτροπή. Εγώ δεν είμαι εμπειρογνώμονας, ούτε έχω χρόνο να ασχοληθώ με τα κείμενα που υποβάλλουν αυτές οι πόλεις. Ούτε και εσείς αδιάκοοι στον χρόνο, ούτε και κανένας από εμά. Και γι' αυτό αποστέλουμε κάποιους εμπειρογνώμονες, οι οποίοι μαζί με τους άλλους, έχοντας εξετάσει όλα τα κείμενα και τις υποψηφιότητες, αποφασίζουν ποια πόλη θα επιλεχθεί από τη χώρα Χ. Και εμεί δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Θα μας υποβληθεί βέβαια κα, καθοδόν. Α, δεν θα χρειαζόταν, αλλά εντάξει, είναι πιο ευγενικό. Είναι μια χειρονομία προ εμά, γιατί και εμείς έχουμε αποστείλει δύο Αλλά και η Κομισιόν δεν αποφασίζει μόνη της. Και το Συμβούλιο δεν αποφασίζει. Η Κριτική Επιτροπή αποφασίζει η οποία αποτελείται από υπερογνώμονες που δεν είσαι ούτε εσύ, ούτε εγώ, ούτε κανένας εδώ, εκτός από τους τρεις εκεί πέρα. Αυτό δεν θα αλλάξει τίποτα. Αλλά σας είπα, το δικαίωμα είναι για μια χώρα να έχει την πολιτιστική πρωτεύουσα, οι προτάσεις δίνονται από τις πόλεις. Καλό είναι. Εάν μια χώρα έχει μόνο μία-δύο υποψηφιότητες, τι να κάνουμε. Αν οι πόλεις δεν ζητούν, δεν μπορούμε να την υποχρεώσουμε. Στο Βέλιο μόνο η Μόντς ήταν υποψήφια. Τι να κάνουμε. Το ίδιο και στο Λουξεμβούργο, ας πούμε. Πού θα βρει κανένας πολύ περισσότερες πόλεις. Mit dem Land nebendran und mit dem, mit dem Land nebendran und mit den anderen Regionen in Κάτι άλλο που θα ήθελα να προτείνω για την πολιτιστική πρωτεύουσα θα πρέπει να σκεφτεί κανένας πώς θα τα οργανώσει Οι γειτονικές χώρες, συνοεύοντες χώρες, πώς θα μπορούν να συνεννοηθούν ίσως. Αλλά το είπε κάτι, κάτι είπαν οι Ότι και άλλα κρατημέρη θα πρέπει να εμφανίζονται στην ε, πολιτιστική πρωτεύουσα είναι σαφές. Πιστεύω ότι στα χέρια της, αν και του προσταμένου και των συναδέλφων βρίσκεται σε καλά χέρια το θέμα. Είναι μια μικρή ομάδα, αλλά αποτελεσματική. Και την άνοιξη του χρόνου νομίζω θα έχουμε μια πρόταση που θα λαμβάνει υπόψη τις προτάσεις που έχουμε υποβάλει και άλλες προτάσεις και θα πρέπει να βελτιώσουμε την πρόταση που μας έχετε υποβάλει. Ευχαριστώ τους εμπειρογνώμονες, ευχαριστώ την Κομισιόν και μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο σημείο της ημερησίας διάταξης. Have a good trip back. So, jetzt haben wir was Schönes. Λοιπόν, έχουμε τώρα κάτι ωραίο. Όχι, αυτό ωραίο ήταν, συγγνώμη. Ε, exchange of views. Έχουμε ανταλλαγή απόψε με τους τρεις βραβευτέντες ε, του βραβείου ε, Καρλομάγνου για την νεολαία. Το βραβείο Καρλομάγνου για την ε, νεολαία είναι νεαρό βραβείο, ιδρύθηκε το 2008. Να τα πείτε κι εσείς. κι εγώ δεν θέλω να μακρηγορήσω γιατί δεν έχουμε και τόσο τρομακτικό αριθμό βουλευτών αλλά ακούνε και οι συνεργάτες και οι βοηθοί τους και είμαστε εδώ για να σας ακούσουμε, να φογκραστούμε αυτό που έχετε να μας πείτε και σας παρακαλώ να πάρετε το λόγο με τη σειρά. Πρώτα, το τρίτο βραβείο. Ο Σουσέ Τούρμο Μαρτίνες, να μας πείτε τι κάνατε, να μας παρουσιάσετε το πρόγραμμά σας σύντομα, περιεκτικά, συστηθείτε. Έχετε PowerPoint θα μας δείξετε τίποτα. the forefront. Ελάτε εδώ μπροστά παρακαλώ. Εσείς έχετε κάτι να παρουσιάσετε. Μάλιστα. Ε, ελάτε μπροστά. Ε, just to tell you how, how... Για να σας πω πώς το κάναμε. In 2011, 240... 245 έργα από τα 27 κράτη-μέλη κατατέθηκαν για το 2011. Ήταν ε, ε, διπλή δύο σταδίων διαδικασία επιλογής, εθνικό σκέλος, ε, δύο ευρωβουλευτές και ένας εκπρόσωπος μιας οργάνωσης νεολαίου ήταν η προεπιλογή και 27 νικητές από τα κράτη-μέλη εκρίθησαν από μια Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τον πρόεδρο Μπούζεκ τον ίδιο τρεις άλλους ευρωβουλευτές και εκπροσώπους ε, του Ιδρύματος Καρλομάγνου και εξέλεξε τους τρεις ε, βραβευθένες αυτή η Επιτροπή, το τρίτο βραβείο λοιπόν ε, και ο λόγος στον κύριο Τόρμο Μαρτίνεθ από την Ισπανία. We have the floor. Come on. Bien, eh, hablaré en español porque estoy seguro. Εγώ θα μιλήσω ισπανικά, γιατί εγώ είμαι σίγουρα ότι οι μεταφράστριες αυτή την αίθουσα τα ξέρουν καλύτερα από μένα. Λοιπόν, εδώ μας αναφέρατε τα σχέδια τα οποία κέρδισαν στον Καρλομάγνιο Νεολαία. Εγώ θα σας παρουσιάσω ένα πρόγραμμα, ένα θεατρικό πρόγραμμα, ε, σχέδιο και ένα σχέδιο έρασμος. Ε, ξέρετε ότι υπάρχουν ένα σωρό Ευρωπαίοι φοιτητές που ζουν για πολλά χρόνια σε άλλες χώρες ανταλλαγές. Εγώ έρχομαι από τη Βαλένσια, ευρωπαϊκή πόλη, από την οποία περνάνε πάνω από 6.000 φοιτητές έρασμου το χρόνο. Εμείς που ανήκουμε στη γενιά του έρασμου είμαστε πεπισμένοι ότι η Ευρώπη έχει νόημα έχει και έχει και πολλά νοήματα. Εγώ έρχομαι να σας μιλήσω εδώ για ένα πολιτιστικό σχέδιο το οποίο θέλει να εκμεταλλευτούμε αυτό το οποίο μας ενώνει και αυτό που μας διαφοροποιεί για να μπορέσουμε να φτιάξουμε την Ευρώπη των ανθρώπων και του πολιτισμού. Στο πρόγραμμα Έρασμος ε, θέλουμε να εκμεταλλευτούμε στα πανεπιστήμια υποδοχής ε, ε, το δυναμικό των νέων που έρχονται και όταν ξεκίνησε το πρόγραμμα Έρασμος, ορισμένοι πίστευαν ότι αυτό το πρόγραμμα θα επέτρεπε απλώς τυπικές ανταλλαγές ε, φοιτητών. Ένας χρόνος σπουδών σε ένα εξωτερικό σε ένα πανεπιστήμιο, μαθαίνεις και μια ξένη γλώσσα, εμπειρία σε μια άλλη πόλη, αλλά είναι αδύνατο να, είχαν φανταστεί κάποιοι τότε ότι σε πολλές ευρωπαϊκές ευρωπαϊκές πόλεις θα δημιουργόντουσαν πολλές μικρές κοινότητες Ευρωπαίων που θα ζούσαν για μία περίοδο σε μια άλλη τρίτη πόλη, σε μία ενιαία κοινότητα. Άλλοι σκέφτονται ότι αυτό είναι λάθος, ότι θα έπρεπε ο έρασμος ε, να εντάσσεται στις πόλεις που τους υποδέχεται και όχι να δημιουργεί παράλληλες πραγματικότητες. Αλλά το ταξίδι αυτών των φοιτητών είναι ένα ταξίδι προς την Ευρώπη και την Ευρώπη αναζητούν όταν ταξιδεύουν. Είτε πρόκειται για την Ισπανία είτε για την Ευρώπη. Ένας φοιτητής του Έρασμου είναι ένας ε, φοιτητής της Ευρώπης και αυτό δεν είναι αλήθεια ότι δεν εντάσσονται στη χώρα υποδοχή. Συμμετέχουν στην πολιτιστική ζωή των πανεπιστημίων και των πόλεων που τους υποδέχονται ε, και γίνονται πρεσβευτές αυτών των χώρων και μαθαίνουν και γλώσσες. Αλλά από την πρώτη μέρα έχουν απόλυτη συνείδηση της εφημερότητας της παραμονής τους μόνο ένα χρόνο. Γι' αυτό προσπαθούν να εκμεταλλευτούν όσο το δυνατόν περισσότερο το χρόνο στην πόλη που τους υποδέχεται, να το βιώσουμε καλύτερα με αυτούς που συμμερίζονται την ίδια κατάσταση με εμά, με τους άλλους εράσμους των άλλων χωρών. Γι' αυτό θα ήταν λάθος για τα πανεπιστήμια και για τις πόλεις υποδοχής να μην εκμεταλλευτούν ε, αυτήν την ιδιαιτερότητα της ε, κοινότητας ε, των Ευρωπαίων φοιτητών που ζουν μαζί μέσα σε μια κοινότητα και έχουν ως χαρακτηριστικό τον φιλοευρωπαϊσμό τους. Ε, πριν από ένα χρόνο ένα αερασιτεχνικό, ένας αερασιτεχνικός θείασος στη Βαλένσια, όλοι πτυχιούχοι, γιατροί, δικηγόροι, μηχανικοί κλπ. Όλοι οι παλιοί ε, φοιτητές. Ε, είπαμε να φτιάξουμε ένα θέατρο. Το θέατρο Έρασμος. Πρόκειται για ένα ευρωπαϊκό σχέδιο με έδρα το Πανεπιστήμιο της Βαλένσια όπου συμμετέχουν φοιτητές Έρασμος δημιουργούνται έτσι θίαση και δίνονται θεατρικές παραστάσεις. Αλλά μέσα ενσωματώνονται όλες οι καλλιτεχνικές δραστηριότητες που απαιτούν ομαδική δουλειά. Ο τελικός μας στόχος είναι να μπορέσουμε να, να έχουμε έναν ε, ε, έρασμο ε, συν network, δηλαδή ένα δίκτυο θειάσεων θεάτρων μάλλον, σκηνών. Και να μπορούμε εκεί να συνενώνουμε την ε, ανθρώπινη εμπειρία ε, και αυτό το, εμείς ε, το παλέψαμε στη Βαλένσια για μερικά χρόνια και είχαμε πολύ σημαντική επιτυχία. Τώρα γιατί ξεκινήσαμε από το θέατρο και θα σας εξηγήσω πώς οργανώνουμε εμείς και τα κούρ στο Πανεπιστήμιο της Βαλένσιας, τα μαθήματα. Empezamos siempre, todos los años, con el Κάθε χρόνο ξεκινάμε εμείς με το θέατρο. Γιατί επιλέγουμε το θέατρο. Γιατί το θέατρο επιτρέπει στους Ευρωπαίους φοιτητές να εργάζονται σκληρά για ένα χρόνο και για να έχουν ένα θετικό τελικό αποτέλεσμα, να ενσωματώνουν όλες τις καλλιτεχνικές ε, ε, τάσεις, όλες τις τους καλλιτεχνικούς κλάδους ε, στο τελικό θέαμα. Υπάρχει, ο, ο κάθε Ευρωπαίος φοιτητής έχει δική του διαφορετική αντίληψη για το θέατρο, διότι αυτό εμπλέκει τη γνώση, τη διάδοση της ευρωπαϊκής κουλτούρας, ε, την επαφή με άλλες ε, κοινοτικές γλώσσες, μας επιτρέπει να δίνουμε αυτή την εμπειρία προς το κοινό και να το μεταφέρουμε αυτό το θέαμα σε άλλα πανεπιστήμια. Εμείς στη Βαλένσια στην αρχή ε, πριν ξεκινήσει το, ε, η περίοδος ε, στέλνουμε πρόσκληση σε όλους τους φοιτητές έρασμος της Βαλένσια εμείς για τα διάφορα ατελειέ έχουμε, συστήνουμε ομάδες 20 ατόμων, το 70% είναι φοιτητές έρασμος και το 30% φοιτητές του Πανεπιστημίου της Βαλένσια. Μέχρι τώρα η, η κοινότητα της Βαλένσια, το Πανεπιστήμιο συγγνώμη, της Βαλένσια χρηματοδότησε τα θεατρικά ατελειέ και ένας ε, καθηγητής ε, είναι αυτός ο οποίος διδάσκει στο πρακτικό, στο ατελείο πρακτικής του θεάτρου. Τα ατελείο θεάτρου στο Πανεπιστήμιο έχουν δύο ε, σκέλη. Ένα πρώτο τμήμα, ένα πρώτο ατελείο το οποίο τελειώνει στα μισά της χρονιάς και όπου δίνουν, οι φοιτητές δίνουν παράσταση του θεάματος που ετοίμασαν και εμείς ε, ε, κάθε φορά για το θέαμά μας ε, επιλέγουμε ένα ευρωπαϊκό θέμα, ένα ευρωπαϊκό σκηνικό, ένα ευρωπαϊκό σενάριο. Αυτό είναι το πρώτο μας θέαμα που κάναμε με φοιτητές από 16 διαφορετικές χώρες. Και εδώ έχετε μία εικόνα το τι κάναμε στην προηγούμενη περίοδο. Και το ατελείε καταλήγει πάντα σε ένα τελικό ε, θέαμα, μια τελική εκδήλωση μας επιτρέπει να παρουσιάσουμε τη δουλειά των πολιτών στην πόλη. Και ε, πήγε αυτή η παράσταση σε 40 διαφορετικά μέλη στην ε, Ισπανία, χωριά, πόλεις. Ε, εμείς κερδίσαμε δύο βραβεία στην Ισπανία για την πολιτιστική μας δράση και μπορέσαμε εμείς να δώσουμε παραστάσεις με 16 διαφορετικούς ηθοποιούς από 16 διαφορετικές χώρες σε φυλακές, σε νοσοκομεία, σε πόλεις, σε χωριά. Σε αυτή την παράσταση έχουμε φοιτητές από 13 χώρες όπου στο ισπανικό κοινό παρουσιάζουν ένα θέαμα ε, με, τις συνήθειε συνήθειες του καθένα. Εδώ έχετε διάφορες εικόνες, έχετε έναν Βούλγαρο φοιτητή με μια Ιταλίδα φοιτήτρια, εδώ έχετε Ιταλούς, Βουλγάρους, Έλληνες και Ισπανούς φοιτητές. Και πέρα από τα θεάματα, οι ίδιοι φοιτητέ οργανώνουν και άλλες δραστηριότητες. Εμείς έχουμε 200 μέλη ε, στην, ε, στο, στο θεατρικό εργαστήρι, στην Βαλένσια, και 100 ε, και πάνω φοιτητές είναι ξένοι. Εδώ έχουμε ένα θέαμα στο δρόμο ε, που παρουσιάστηκε στο φεστιβάλ του θεάτρου το δρόμο, στο δρόμο όπου οι Ευρωπαίοι φοιτητές εξέφρασαν την ανησυχία τους για το πώς εξελίσσεται σήμερα η ιδέα της Ευρώπης. Έχουμε μία μεγάλη, μία ορχήστρα, μία big band ε, και σήμερα ε, φέτος άρχισε να λειτουργεί το Erasmus in Network στο ε, Μαγδεμβούργο, ε, στη Γρανάδα, στην Κρακοβία, στην Μπολόνια, στην Κοπεχάγη. και στη Γαλλία επίσης. Δεν είναι ένα ισπανικό σχέδιο αυτό. Ξεκίνησε από την Ισπανία. Θέλουμε να, να, να συνεχιστεί στην υπόλοιπη Ευρώπη. Στις 29-30 Μαρτίου έχουμε μία συνάντηση στην Ισπανία, ούτως ώστε αυτή η σκηνή, αυτό το θέατρο Εράσμους ε, να επεκταθεί στην υπόλοιπη Ευρώπη, να κάνουν όλοι οι υπόλοιποι αυτό που κάναμε στη Βαλένθια. Θέλουμε μία δομή Θέλουμε μία διαδρομή ούτως ώστε να υπάρχει ορατότητα για τις πολιτιστικές εμπειρίες όπου συμμετέχουν οι νέοι Ευρωπαίοι, οι νέοι φοιτητές. Θέλουμε να έχουμε ανταλλαγή μεταξύ των πανεπιστημίων της Ευρώπης και να περάσουμε πέρα από αυτό, να κάνουμε ένα βήμα παραπάνω, να έχουμε ένα βήμα μεγαλύτερο προς την Ευρώπη. και να μπορέσουμε να ε, προβάλλουμε και άλλες μορφές ε, τέχνης, ε, την μουσική ή τις οικαστικές τέχνες. Θα θέλαμε λοιπόν εμείς να εκμεταλλευτούμε όλο αυτό το δυναμικό, το, το, το, το, πολιτιστικό και ανθρώπινο δυναμικό των Ευρωπαίων φοιτητών για να μπορέσουμε να οικοδομήσουμε μια Ευρώπη του πολιτισμού και των προσώπων, μια Ευρώπη που εμείς θεωρούμε ότι θα πρέπει να είναι ορατή σε όλες τις χώρες, σε όλες τις πόλεις. Μια θετική Ευρώπη που θα μπορούσε να φωτίσει αυτήν την άλλη Ευρώπη που μας ε, απαγοητεύει τόσο πολύ σήμερα που είναι η Ευρώπη των αγορών και του νομίσματος. Γι' αυτό λοιπόν ε, θα θέλαμε για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε να έχουμε την υποστήριξή σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, σας ευχαριστώ κύριε Μαρτινές. Είναι καταπληκτικό αυτό που έκανε και ελπίζω να έχετε πολλή επιτυχία και πολλή δικτύωση και σε άλλες πανεπιστήμιοι πόλεις. Γιατί αυτή η ιδέα πραγματικά προωθεί την Ευρώπη κάτω από ένα διαφορετικό φως. Ιδίως στην εποχή κρίσης που χρειαζόμαστε το φως στην άκρη του τούνελ. Συνεχίστε έτσι τώρα. Θα ήθελα να δώσω το ρόλο στον Κωνσταντίνο Ταντίνο που έχει το δεύτερο 10 λεπτά, έτσι. Ναι, σας ευχαριστώ για την ε, πρόσκληση. Ε, Βαλκάνια πέρα των συνόρων είναι μια μη κυβερνητική οργάνωση που βασίζεται αυτή τη στιγμή στο Αθήνα. Δημιουργήθηκε στο Βερολίνο όπου πέντε άτομα αποφάσισαν να δημιουργήσουν ένα φεστιβάλ κινηματογράφου για να μπορέσουν να προωθήσουν την ιδέα αυτή μεταξύ των νέων στα Βαλκάνια. Πιστεύουν ότι το φεστιβάλ αυτό θα μπορούσε να είναι ένα σημείο συνάντησης των νέων της περιοχής. Η οργάνωση αυτή ε, οργανώνεται από εννέα επαγγελματίες, ε, κυρίως από τις χώρες των Βαλκανίων, τα Δυτικά Βαλκάνια, που γνωρίζετε εσείς πολύ καλά κυρία Πακ. Ο στόχος μας είναι να δημιουργηθεί η συνεργασία μεταξύ των νέων και δεύτερον να προωθεί η ευρωπαϊκή ιδέα στον, ε, στην περιοχή χρησιμοποιώντας ήχο και εικόνα. Ε, εμείς ε, προωθούμε την πολιτιστική πολυμορφία της περιοχής τονίνοντας ε, την ε, τον βαλκανικό πολιτισμός προωθώντας και την κινητικότητα των νέων. Ο στόχος είναι να καλέσουμε όλους να συμμετάσχουν στη δική μας δραστηριότητα αλλά να οργανώσουν και δικές τους τοπικές δραστηριότητες. Επίσης προσπαθούμε να προωθήσουμε το διάλογο και συνεργασία μεταξύ νεολαία σήμερα για ένα καλύτερο αύριο. Τα Βαλκάνια χωρίς σύνορα ε, δημιουργούν μια μορφή έκφρασης ε, για τους νέους, ε, μια πλατφόρμα για να μπορέσουν να γνωρίσουν την βαλκανική πολιτιστική πτυχή πετυχαίνουμε τους στόχους μας με τέσσερους ε, τρόπους. Με ένα φεστιβάλ ε, φιλμ, τα εργαστήρια, τα σεμινάρια και το ε, διαβαλκανικό δίκτυο. Όπως είπα και προηγουμένως, χρησιμοποιούμε κυρίως εικόνα και ήχο. Η κύρια μας λοιπόν δραστηριότητα είναι το φεστιβάλ που οργανώνεται κάθε χρόνο σε διαφορετικές χώρες των Βαλκανίων. Το 2010 ήταν στο Βελιγράδι με το θέμα συνεργασία στα Βαλκάνια. Το 2011 Αθήνα. Ποιο ε, φοβάται τη μεγάλη κακή κρίση. Ήμασταν εκεί κατά τη διάρκεια της κρίσης ε, το Ιούνιο. Του χρόνου θα έχουμε στα τύρανά το θέμα «Μίλησέ μου». Πολυγλωσία και επικοινωνία. Και σας καλούμε να έρθετε. Αλλά η επιτυχία αυτού του φεστιβάλ μας οδήγησε και σε άλλες δραστηριότητες για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε με τους στόχους μας. Ε, οργανώσαμε κάποια ακαδημαϊκά σεμινάρια με πιο ακαδημαϊκή ε, προσανατολισμό, όπου ο στόχος μας ήταν οι πρωτοετής φοιτητές, όπου είδαμε ότι δεν γνωρίζουν καθόλου τις γειτονικές χώρες στην περιοχή. Ε, ασχολούνται με τις ανησυχίες της ε, περιοχής και παρουσιάζεται μια μικρή ταινία που είτε πα, δημιουργείται κατά τη διάρκεια των ε, εργαστηρίων ή είναι εκείνη που είχαμε στο φεστιβάλ. Επίση έχουμε εργαστήρια που νομίζουμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για την συνεργασία, την κοινή συνεργασία να συνοθούν νέοι από διάφορε χώρε τη ε, Νοτιοανατολική Ευρώπη για να συζητήσουν και να έχουμε θετικέ εμπειρίες. Το 2011 είχαμε τρία ε, εργαστήρια, το ένα στα Σκόπια, το άλλο στα Τίνιρανά και το τρίτο στην Αθήνα πάλι με το θέμα ποιος φοβάται τη μεγάλη κακή αυτή κρίση. Πάντα τα εργαστήρια αυτά έχουν το ίδιο θέμα και συνενώνουν μια σειρά δραστηριοτήτων. Και τέλος, όπως είδαμε όλοι, ότι είναι σημαντικό το δίκτυο για προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα δίκτυο στα Βαλκάνια, ένα δίκτυο που όσο πάει και τόσο πιο ε, διευρύνεται στην περιφέρεια και προσπαθούμε να εμπλέξουμε κατά δυνατόν πολλούς νέους επαγγελματίες στην περιοχή. Και γι' αυτό έχουμε την έννοια των ε, πρέσβειων BBB. Προσπαθούμε δηλαδή έτσι να προσφέρουμε ένα πλαίσιο για να γνωριστούμε, να κάνουμε φίλους και βλέπουμε τι λειτουργεί το θέμα. Πιστεύω, όπω είπε και ο Μαξ Φερότ, εκείνο που γνωρίζει έναν δεν ξέρει κανέναν. Είναι αληθέ. Μπορείτε να μας βρείτε στο facebook, στο twitter, παντού ακολουθούμε αυτά τα νέα μέσα. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σα και σας ευχαριστώ που μας δώσετε τη δυνατότητα να είμαστε εδώ. It's clear that you are... Ευχαριστώ πολύ. Προφανώς είστε στο facebook και αν δεν είστε να μπείτε εσείς από τον έρασμο. Ακολουθήστε αυτό το δρόμο, λίμωνο. Πολύ καλή ιδέα επίσης και προσωπικά με συγκινεί γιατί είμαι πολύ προσιλωμένη και δεσμευμένη και αγωνίζομαι για τα Δυτικά Βαλκάνια και την Νότιο-Ανατολική Ευρώπη. Τώρα έχω και το χαρτί μου. Ο πρώτο βραβευτή είναι από το Ηνωμένο Βασίλειο, την πιο φιλοευρωπαϊκή χώρα όλων των εποχών. Έχετε το λόγο, κύριε Σύρμα. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα μιλήσω αγγλικά, ζητώ συγγνώμη από του διερμηνεί εκ των προτέρων. Η Ευρώπη και εγώ είναι ένα δικτυακό επιγραμμικό περιοδικό που δημιουργήθηκε από νέους Ευρωπαίους για νέους Ευρωπαίους τελείως εθελοντικά λειτουργεί για να είναι η Ευρώπη πιο προσωπική. Γιατί θεωρούμε ότι η Ευρώπη ε, ταυτίζεται μόνο με τη γραφειοκρατία και αν γίνει αυτό και με τις Βρυξέλλες οι νέοι Ευρωπαίοι δεν θα μπορούν να ταυτιστούν με αυτοί. Εμείς το κάνουμε με ένα τριμηνίο περιοδικό και έχουμε και ε, Facebook και Twitter και εργαστήρια. 9 εκδότες από 7 διαφορετικές χώρες και 100 συντάκτες από όλες τις χώρες της Ευρώπης. Η διεθνής η προσπάθεια ε, για την ευρωπαϊκή ε, δημοσιογραφία. Μπορείτε να το δείτε στην ιστοσελίδα μας. Να σας πω τι κάναμε σε τέσσερα χρόνια. Μάλλον σε τέσσερα χρόνια τι θα γίνει. Το 2015 δεν θα είναι μόνο στην πρωτοπορία το ε, περιοδικό, αλλά θα εκπαιδεύει και νέους δημοσιογράφους. Ε, μια διεθνική εγκάρσια προσέγγιση για την Ευρώπη. Τι εννοώ και τι σημαίνει. Δεν περιορίζονται από εθνικά συμφέροντα τα άρθρα μας, αλλά, όπως κάνουν κάποια κοινωνικά δίκτυα, αλλά θέλουμε να καταλάβουμε τι είναι η Ευρώπη και πώς αλλάζει η Ευρώπη. Γιατί η Ευρώπη δεν ορίζεται από τα θεσμικά όργανα της. Η Ευρώπη είναι τρόπος σκέψης, είναι νοοτροπία, είναι κόσμο θεωρία. Είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τον κόσμο. Και ε, οι νέοι επαγγελματίες μπορούν να αναπτύξουν εκεί την εργασία τους και να περάσουν ε, την Ευρώπη σε μια νέα διάσταση. Ε, εκπαιδεύουμε δημοσιογράφους που επιστρέφουν στα κλασικά μέσα ενημέρωσης και βλέπουν τι γίνεται με την Ευρώπη και θα δημιουργηθεί ένας πραγματικά δημόσιος χώρος. Σε τέσσερα χρόνια από σήμερα θα έχουμε και υποστήριξη και δημόσια και ιδιωτική. Επί δύο χρόνια είχαμε ε, ένα με δύο εργαζομένους πλήρους απασχόλησης και έχουμε ε, ήδη εθελοντική εργασία ε, για να πετύχει το πρόγραμμα του χρόνου. Θα είμαστε στη δράση 4,5 Καταλαβαίνετε ότι κερδίσαμε το βραβείο Καρλομάγ με καμία οικονομική υποστήριξη και δημιουργήσαμε ένα περιοδικό και ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης νέων δημοσιογράφων. Κοιτάξτε για μας τι σημαίνει Ευρώπη. Θα το καταλάβετε με αυτό το διάγραμμα. Έχουμε λοιπόν ένα πρόσωπο ε, με ε, έναν άνθρωπο με τον εγκέφαλο που είναι ε, η σκέψη, η Ευρώπη των πολιτικών, την καρδιά στη συνέχεια, ε, το διάφραγμα, την κοιλιά που κυοφορούνται τα βρέφη στην Ευρώπη και τα πόδια που είναι για το περπάτημα, πώς τα πού πηγαίνει η Ευρώπη. Αυτές όλες είναι οι κατηγορίες που αφορούν την Ευρώπη και εμένα. Το blog που είναι η πλατφόρμα η δική μου ονομάζεται έκτη αίσθηση και θέλουμε πραγματικά να κάνουμε τον ευρωπαϊκό ε, τύπο ή την ε, δημοσιογραφία, ε, την ευρωπαϊκή ουσιαστική και πραγματική. Γράφει ένας Πολωνός για τις πολωνικές εκλογές και δείχνει πώς η ευρωπαϊκή συζήτηση επηρεάζει τις πολωνικές εκλογές και πώς οι πολωνικές εκλογές με τη σειρά τους επηρεάζουν την υπόλοιπη Ευρώπη. Εκτός από το περιοδικό έχουμε και τρία μεγάλα έργα φέτος. Να σας εξηγήσω σύντομα τι κάναμε και γιατί το κάνουμε αυτό. Πρώτον, ε, ένα ατελιέ εργαστήρι τον Ιανουάριο σε συνεργασία με ένα Ινστιτούτο για εκπαίδευση νέων δημοσιογράφων ε, με εκθέσεις ιδεών ε, για το πώς αντιλαμβάνονται την Ευρώπη. 20 υποψηφιότητες ήρθαν για την πρώτη φορά. Πώς αντιλαμβάνομαι την Ευρώπη και τι σημαίνει για μένα η Ευρώπη. Το Δεκέμβριο με άλλους τρεις φορείς θα διοργανώσουμε ένα εργαστήρι με τίτλο «Μιλάτε Ευρωπαϊκά». Αυτό έχει να κάνει και με ε, τη δημοσιογραφία και με τη μουσική και με τις πεπιθήσεις. Για πρώτη φορά συμμετέχουν Ρουμάνοι. 650 ήταν υποψηφιότητες για 25 θέσεις και μόνο. Και όλα αυτά ε, αποκρισταλώνονται σε μια μόνιμη πλατφόρμα στην ιστοσελίδα. Δεν είναι απλό περιοδικό. Συμμετέχουν, συνεργάζονται νέοι που θεωρούν ότι είναι υπόθεσή τους η Ευρώπη. Επίσης, έχουμε και ένα debate για την Ευρώπη. Συμμετέχουν νέοι Ευρωπαίοι και ε, συζητούν. Εδώ δεξιά βλέπετε το ε, Ιωάννης ε, που είναι ένας δικός μας και αριστερά ο Άντριαν, ένας υποψήφιος που έχει γράψει ε, ένα άρθρο για την ε, μάχη με δημοσιογραφία. Και το τελευταίο σχέδιο. Συνεργαζόμαστε στο Βερολίνο με το Υπουργείο Εξωτερικών της Γερμανίας για την εξωτερική πολιτική του Βερολίνου. Και ψάξαμε να δούμε πώς βλέπουν την εξωτερική πολιτική και την ευρωπαϊκή πολιτική εν γέννη οι νέοι Ευρωπαίοι. Οχτώ εθελοντές συμμετείχαν και εγώ μαζί και κάναμε μια έρευνα μεταξύ 6.500 Ευρωπαίων. Αυτό είναι εξαπλάσια μελέτη από ό,τι έχει γίνει συνήθως. Και σας λέω τα αποτελέσματα ε, σε ένα γράφημα που είναι βεβαίως ε, προσωρινά. Το πρώτο ήταν αισθάνεστε ότι είστε ενημεροί για τα θέματα της ευρωπαϊκής πολιτικής και εξωτερικής πολιτικής. 2.000 είπανε ναι, και 4.000 είπαν όχι, διπλάσιοι. Γιατί όμω είπαν όχι και μα ενδιαφέρει αυτό να το μελετήσουμε. Αυτό το βλέπετε, ότι δεν μα εξηγούν τα μέσα ενημέρωση. Αυτή ήταν η πιο δημοφιλή απάντηση. Γι' αυτό κάναμε και αυτό το περιοδικό. Εμείς εξηγούμε γιατί καθιστούμε τα ευρωπαϊκά θέματα προσωπικά και τα παρουσιάζουμε με έναν τρόπο που προσελκύουν τους νέους. Ε, ε, γενικό δεν υπήρχε μέχρι τέτοιο πλαίσιο μέχρι σήμερα. Έχουμε δύο εκπροσώπους που πήγαν ε, στο γερμανικό, ελληνικό και πολωνικό Υπουργείο Εξωτερικών, ε, εγώ και ένας συνάδελφός μου, για να παρουσιάσουν αυτές τις ε, απαντήσεις της δημοσκόπησης. Πραγματικά δεν θέλουμε να εργαζόμαστε απομονωμένα, εργαζόμαστε σε συνεργασία και με άλλους φορείς. Εμείς είμαστε για το Ευρωπαϊκό Έτος Εθελοντισμού ε, συνομιλητής επίσημος φορέας και όπως είπε ο πρόεδρος Μπούζεκ όταν μας απένιμε το βραβείο η Ευρώπη ε, είναι ένα σχέδιο και αυτό που θέλουμε είναι να κάνουμε την ευρωπαϊκή ιδέα ελκυστική cool τώρα που ο κόσμος αναδιπλώνεται στα εθνικά του πλαίσια και φοβάται Θέλουμε εμείς η Ευρώπη να μην συνδέεται με τη γραφειοκρατία και τη διοίκηση. Οι νέοι Ευρωπαίοι θα πρέπει να συνδέουν την Ευρώπη με την εμπειρία τους, με ένα lifestyle και να ταυτίζονται με την Ευρώπη, να γίνεται πιο προσωπική και να εκπαιδεύσουμε μια νέα γενιά δημοσιογράφων πέρα από τα εθνικά σύνορα, διεθνή. Μόνο έτσι θα έρθει και ο ευρωπαϊκός πολιτισμός κοντά σε ανθρώπους που ποτέ δεν θα τους έφτανε. Στόχος μας είναι να περάσουμε σε ένα επόμενο επίπεδο οι νέοι Ευρωπαίοι να μάθουν την Ευρώπη, να εκπαιδευτούν διαβίου και η Ευρώπη να είναι προσωπική, να συμπεριλαμβάνει τους νέους και ε, πανευρωπαϊκή. Εξ ονόματος ε, των συντακτών και των εργαζομένων στο περιοδικό αυτό, σας ευχαριστώ πολύ. Thank you very much. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ κύριε Σέρμαν. Εντυπωσιακά όλα αυτά, πάρα πολύ. Ελπίζω επίσης πάρα πολύ να έχετε και πολλούς ε, που να σας παρακολουθούν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Γιατί είναι πολύ επικίνδυνο. Τουλάχιστον τρία γερμανικά ιδρύματα σας χρηματοδοτούν και αυτό είναι πάρα πολύ ύποπτο. Προσοχή. Προσέξτε. Μερικοί θα πούν ότι είναι εισβολή γερμανική, Ηνωμένο Βασίλειο, κάμια τέτοια εισβολή. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ όλους σας. Εγώ θέλω να σας φίξω όλους στην αγκαλιά μου, γιατί ε, θεωρώ ότι χρειαζόμαστε ανθρώπους σαν και εσάς. Έχετε έρθει εδώ και πολλοί άλλοι ε, που ε, υπέβαλαν υποψηφιότητα. Είναι πολύ λίγες οι δυνατότητε μόνο, είναι πολύ λίγα τα χρήματα. Τρεις από εσά μόνο βραβεύεστε. Τα πήρατε τώρα, ελπίζω να πιάσουν τόπο σε καλή μεριά και σα αφαιρύνουμε να προχωρήσετε. Εδώ έχουμε και τέσσερις του ΕΛΚ, μία πράσινη βουλευτή και έναν της αριστεράς. Για να καταλάβετε λίγο πώς έχουν τα πράγματα. Όλοι οι άλλοι είναι βοηθοί, συνεργάτες διαφόρων πολιτικών ομάδων. Είναι πολύ εύκολο όλα αυτά, έτσι δεν είναι. Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Σταματάω τώρα τα γλυκούλια μου και τα εσπεράντο. Σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε ε, ε, Καλή σας επάνωδο, ό,τι επιθυμείτε, συνεχίστε την προσπάθειά σας. Ερχόμαστε στο σημείο 13, αποφάσεις των συντονιστών τις έχετε λάβει όλοι. 14 διάφορα, δεν έχουμε τίποτα, 15, 22, 23 του μηνός επόμενη συνεδρίαση. Ευχαριστώ τους διερμηνείς και σας εύχομαι καλό βράδυ. Γεια σας.